Meine Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Δεν έχουν έρθει ακόμα πολλοί συνάδελφοι. Ωστόσο πρέπει να ξεκινήσουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διότι έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα. Επειδή δεν θέλουμε να συνεχιστεί η συζήτηση και την Τετάρτη το απόγευμα, θα ήθελα να προχωρήσουμε γρήγορα. Δύο παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, όπως ε, βλέπετε δίπλα μου δεν κάθεται ο Υπουργός Φελίτζη, αλλά ο Ιβαν Κόβατς, που είναι αναπληρωτής ε, υφυπουργός, τον οποίο έχουμε γνωρίσει και σε άλλες περιστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να τον καλωσορίσω και θα έχουμε συζήτηση μαζί του στο θέμα υπαρθμών 4 της ε, διάταξη. διάταξης. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν και παρακαλώ να πείτε περαστικά στον Υπουργό από μας. Δεύτερη παρατήρηση. Την Τρίτη στις 4 ε, η ώρα το απόγευμα έχουμε μια τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη θα έρθει ο κύριος Τάνακα. Ε, έτσι λοιπόν θα έχουμε αλλαγή στη σειρά της ημερησίας διάταξης. Ήθελα να το... Ήθελα να ενημερωθούν οι συνάδελφοι διότι ε, η γραμματεία δεν το, έκανα. Δεν, το, δεν το έκανε. Και έτσι θα έχουμε το ΚΚΠ ω θέμα υπαριθμών 18 στην ημερησία διάταξη. Και η έκθεση θα πάει μετά τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα γίνει ένα σεμινάριο του Τμήματος Πολιτικής ε, για το θέμα της διαστημικής τεχνολογίας που θα στηρίξει την ευρωπαϊκή πολιτική την Τετάρτη το απόγευμα. Το γνωρίζουν όλοι νομίζω, απλά ήθελα να σας, πω, να σας θυμίσω ότι είμαστε υπεύθυνοι για τη διαστημική πολιτική μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, μπορεί λοιπόν να σας ενδιαφέρει να περάσετε να ακούσετε την συζήτηση. Και επίσης θα μας εγκαταλείψουν δύο μέλη της γραμματείας ε, και ήθελα να πω δύο λόγια, αλλά δεν είναι παρόντες από ό,τι βλέπω. Ωραία. Να σας πω ότι κατά τα άλλα έχουμε τα πρακτικά. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουν εγκριθεί και προχωράμε στο ε, σημείο 4 και θα ήθελα να καλωσορίσω και πάλι τον κύριο Κόβατς. Θα θέλαμε να εξετάσουμε τα αποτελέσματα της Ουγγρικής ε, Προεδρίας ε, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ ταραγμένες εποχές. Και παρότι ήταν ταραγμένε εποχέ και υπήρχαν πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη τα οποία δεν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων, ε, νομίζω ότι καταφέραμε αρκετά ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή μα. Ε, Σα δίνω το λόγο λοιπόν, παρακαλώ. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, it's good to be here.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 különösen a fő Hangsúlyt kell fektetnünk azokra a szektorokra, amelyekben a legnagyobb energia megtakarítási pot. Θα πρέπει επίση να εστιάσουμε στου τομεί αυτού όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονομήσεων και εδώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στι μεταφορέ και στην κατασκευαστική βιομηχανία. Ο δημόσιο τομέα εδώ έχει να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο, παραδείγματο χάρη μέσω των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, μέσω επενδυτικών κινήτρων, μέσω κανονισμών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Επέκεινα τώρα όλων αυτών των στοιχείων της στρατηγικής υπάρχει και μία ακόμα, η, μία ακόμα περιοχή που θέλουμε να δράσουμε και έχει να κάνει με την διαφάνεια των αγορών ενέργειας. Στις 10 Ιανουαρίου 2010 η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση στο Συμβούλιο με νομικές ρυθμίσεις που είναι κατά κάποιο τρόπο μια απάντηση στην χρηματοπιστωτική κρίση. Εξετάζοντας τις αγορές η Κομισιόν ήθελε να ενισχύσει την αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου, το εμπόριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την διαφάνεια, την ε, διάδοση πληροφοριών. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν ρυθμίζονται από το νομοθέτημα αυτό. Έχουμε κάνει συζητήσει για τα θέματα αυτά που πήγανε πολύ καλά. Χάρη και στον Γιώργο Χατζημαρκάκη, τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μα για τα θέματα αυτά. <clears throat> Και στι 2 Ιουνίου μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στι τριγωνικέ ε, συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πετύχαμε λοιπόν περισσότερο από αυτά που ελπίζαμε να πετύχουμε και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Επιτροπή σας για την συμβολή σας. Ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε και τις αποφάσεις αυτές όταν, από ό,τι γνωρίζω, θα ψηφίσετε αύριο για το θέμα αυτό. Ως συμπέρασμα τώρα, ως κατακλείδα, θα ήθελα να σταθώ στα θέματα τα κλιματικά ε, έχουμε τη διασυψη κορυφή του Ντάρμπον που θα γίνει στο τέλο του 2011. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολήσει. Επίση και το τι θα γίνει μετά το 2012. Η Ουγγρική Προεδρία έχει κάνει έχει διοργανώσει στρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίε. Ο στόχο μα είναι να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο είναι φιλόδοξο και νομικά δεσμευτικό ω θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή θέση για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λαμβάνοντα υπόψη το μέλλον του πρωτοκόλου του Κιώτο. 4 Μαρτίου κάναμε μια σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος, όπου το Συμβούλιο κατέληξε σε μια σειρά συμπερασμάτων. στι 24 και 26 Μαρτίου επίση υπήρξε και μια άτυπη σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος και στι 21 ε, Ιουνίου άλλη μία σύνοδο των Υπουργών περιβάλλοντο για να δουν το έργο των ομάδων εργασία και να συζητήσουν σε πολιτικό επίπεδο για την πρόοδο τη ομάδα τη εργασία. Θέλουμε επίσης να ακολουθήσουμε και ένα οδηγό χάρτη για τη μείωση της χρήσης άνθρακος στον ενεργειακό τομέα. Ο στόχος μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση και εκπομπή άνθρακα και θέλουμε να θεσπίσουμε μια σειρά στόχων μέχρι το 2050. Είναι μια νέα και σημαντική στρατηγική στην οποία θέλουμε να συμπεριλάβουμε πολλούς οικονομικούς τομείς. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να συνδέσουμε όλα αυτά με, την, ε, με τον οδικό χάρτη και τις προσπάθειές μας για την απόδοση, την ενεργειακή απόδοση. Πρέπει φυσικά να σκεφτούμε και τις επενδύσεις και να προωθήσουμε την έρευνα για να προχωρήσουμε την ατζέντα αυτή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμα, γι' αυτό θέλω να σας πληροφορήσω από την πλευρά της Ουγγρικής Προεδρίας ότι συζητήσαμε ήδη σε επίπεδο εμπειρογνώμων και σε επίπεδο υπουργών για τα θέματα αυτά. 24 και 26 Μαρτίου, όπως σας είπα, ήταν η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Περιβάντος κοίταξαν μια σειρά θεμάτων, κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα, παρέπεμψαν και στο Συμβούλιο στις 21 <clears throat> Ιουνίου μια σειρά συμπερασμάτων και αν μπορώ τώρα να κλείσω κυρίε και κύριοι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα κρατημέλη και την Κομισιόν και εσάς ως μέλη του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χάρη σε εσά και μόνο χάρη σε εσά μπορέσαμε να επιτύχουμε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας μα. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξη που δώσατε στο πρόγραμμα τη Ουγγρικής Προεδρία και στου στόχου μα και σα ευχαριστώ για την εξασφάλιση τη επιτυχία της Ουγγρικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ και για την προσοχή σα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύψατε και δίνω τώρα το λόγο στους ομιλητές, πρώτα στον κύριο Γκιόρκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Φυπουργέ. Δεν θέλω ακριβώ να σα ε, θέσω μια ερώτηση. Θα ήθελα όμω να σα ευχαριστήσω και να σα συγχαρώ. Να σα ευχαριστήσω για τη συνεργασία ανάμεσα στην Ουγγρική Προεδρία και το Κοινοβούλιο. Η Ουγγρική Προεδρία μα είχε υποσχεθεί ότι θα φερθεί φιλικά απέναντι στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μα ε, και ε, από ό,τι μπορώ να κρίνω εγώ, ε, έχετε εκπληρώσει αυτή την υποσχεσή σα. Αναφερθήκατε στο Ρέμιτ ε, καμιά δύο φορέ. Είμαι σκιώδη συζητή του ΕΛΚ για το θέμα αυτό και γι' αυτό είχα τη δυνατότητα να εξετάσω το φάκελο αυτόν και να εδώ ε, τι σχέσει ε, Προεδρίας ε, και Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στον τριμερή διάλογο. Πόσο φιλικοί ήσασταν απέναντί μας. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία για τη δουλειά της πάνω στο θέμα αυτό. Και όπως είπα, η Ουγγρική Προεδρία ήταν πολύ θετικά διακείμενη απέναντι στο Κοινοβούλιο. Ήδη έχουμε μπει στην Πολωνική Προεδρία, αλλά βρίσκεστε ακόμα εδώ σήμερα στην αίθουσα. σα ευχαριστώ λοιπόν που βρίσκεστε εδώ. Σας συγχαίρω λοιπόν και πάλι για τα όσα επιτύχατε. Πιο ισχυρή Ευρώπη ήταν ένα από τα συνθήματα τη ε, Ουγγρική Προεδρία. Ε, το αναφέρατε αυτό στην αρχή τη ομιλία σα ε, και στον τομέα τη ενεργειακή πολιτική. Νομίζω ότι αναμφίβολα έχετε πετύχει προόδου προ μια πιο δυνατή και πιο ενωμένη Ευρώπη. Νομίζω ότι είμαστε πιο ισχυροί από ότι ήμασταν πριν από ένα εξάμεινο και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ενέργεια αποτέλεσε σημαντική επιτυχία ξεφύγαμε από τα λόγια, έχουμε προχωρήσει πια στις πράξεις και αυτό είναι πολύ θετικό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις ε, αποφάσεις ε, που ελήφθησαν κατά τη συνάντηση κορυφής. Ε, δύο προκλήσεις είχε να αντιμετωπίσει η Προεδρία. Καταρχήν την εφαρμογή του δικού σας προγράμματος και δεύτερον είχατε και τις αναπάντηχες εξελίξεις τις οποίες δεν, μπορούσατε να γνωρίσετε εκ των προτέρων. Εργαστήκατε όμως πολύ σκληρά και νομίζω ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειά. Για παράδειγμα, τα όσα έγιναν στην Βόρεια Αφρική, αλλά και τα stress test ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη ενέργεια. Ε, νομίζω ότι έχετε πετύχει σημαντικέ πρόοδου στο θέμα αυτό. Κανεί δεν το, μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Όσον αφορά το δικό σα ε, πρόγραμμα, ήταν φιλόδοξο και νομίζω ότι αυτό ήταν πρόκληση από μόνο του. Ε, και πάλι όμως ε, είχατε πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Όσον αφορά την ενιαία αγορά ενέργειας και το REMIT, επιτρέψτε μου να πω κανένα δύο λόγια. Ε, αυτά που έχω να πω δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με το, το περασμένο εξάμεινο, πιο πολύ αφορούν το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να πω λίγα λόγια. Έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε ε, ε, πέρα από την αρχική ανακοίνωση της Κομισιόν. Έχουμε το ε, ενιαίο πρόγραμμα, σύστημα καταχώρησης. Έχουμε επίσης την διαβίβαση δεδομένων για το διοξείδιο του άνθρακα στους ενδιαφερομένους και έχουμε και τις κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλονται στο μέλλον. Και αυτό είναι σημαντικό βήμα. Καταφέραμε λοιπόν να πετύχουμε κάποια συμφωνία, τουλάχιστον όσον αφορά τους στόχους. Το επικροτώ αυτό. Και κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση. Πώς βλέπετε το μέλλον, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα πετύχουμε τους στόχους αυτού στην πράξη. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ πλήρης η παρουσίαση που κάνατε έχετε καλύψει τόσες πολλές δράσεις, τόσες πολλές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ουγγρική Προεδρία. Έχω δύο ερωτήματα προς εμάς. Το πρώτο ερώτημα είναι για την ενεργειακή πολιτική που ακολούθησε η Ουγγρική Προεδρία. Ποια είναι η δράση για την οποία είσαστε πιο υπερήφανος. Τι ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα λοιπόν της Ουγγρικής Προεδρίας το εξάμεινο αυτό. Και το δεύτερο ερώτημά μου τι θα συνιστούσατε στην Πολωνική Προεδρία να ακολουθήσει μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε να ακολουθήσει και αυτή η μεγάλη το ένα δρόμο επιτυχίας για τα ενεργειακά θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για τις πληροφορίες που μας παρουσίασε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατήρησεις και κάποιες ερωτήσεις. Τονίσατε ότι είναι για την Ουγγρική Προεδρία υπήρξε η ενεργειακή απόδοση μία από τις προτεραιότητές σας και επίσης και η, η οδηγία για την διαφάνεια της αγοράς ενέργειας ήταν ένα από τα σημαντικά θέματα που σας απασχόλησε. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία μπόρεσατε να έχετε, είσαστε ικανοποιημένοι για τα νομοθετήματα αυτά. Και επίσης θα ήθελα να θέσω το ερώτημα τι πρόοδο έχετε επιτύχει σε σχέση με τον Ναμπούκο. Αν αυτό είναι πράγματι για σας, υπήρξε για σας πράγματι μια, μια προτεραιότητα στον ενεργειακό χώρο και αν όλα αυτά συνάδουν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο που ζήτησε να υπάρχουν καλύτερες διασυνδέσεις στον ενεργειακό τομέα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να υπάρξει μια καλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα σήμαινε ότι θα είχε μεγάλη σημασία ο νότιος διάδρομος και συγκεκριμένα ο Ναμπούκο. Και κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια επιτάχυνση της εφαρμογής του σχεδίου Ναμπούκο γιατί προχωρά χελονοειδώς μέχρι στιγμής και θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι έχετε πράξει για τα θέματα αυτά και τι βλέπετε να ήταν τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. <clears throat> Επίσης, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα κατά πόσο η έκθεση της Κομισιόν που θα δοθεί στο τέλος του θα έπρεπε να είχε δοθεί μάλλον στο τέλος Ιουνίου του 2011 σε σχέση με τις ανάγκες επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. Δεν ξέρω αν έχετε λάβει αυτή την έκθεση από την Κομισιόν και εάν ναι, ποια είναι τα επόμενα βήματα στα οποία προτίθεται το Συμβούλιο να προβεί, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας. Και ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την απόδοση, την ενεργειακή απόδοση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση έχει γίνει δεκτή και περιλαμβάνει συγκεκριμένου και φιλόδοξου στόχου ιδίω σε ό,τι αφορά τα κτίρια, την κατανάλωση ενέργεια στα κτίρια. Ω εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την αποδοτική, ενεργειακή συγγνώμη, απόδοση των κτιρίων, εγώ έχω θεωρήσει ότι ο μηχανισμός ευκαμψίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. Εμείς είχαμε ζητήσει μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο προτείνετε εσείς για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τι μέτρα έχετε λάβει ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μια μεγαλύτερη ευκαμψία μέχρι 15% στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή και εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί το 15% να εξασφαλιστεί τουλάχιστον ένα ελάχιστο κατόφλι 10% για την αύξηση ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Κυρία Καρβάλιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία. Ήταν έξοχο το έργο που επετέλεσε και άριστη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τι προσδοκίες έχετε για τη διάσκεψη του Ντέρμπαν. Πλησιάζει το τέλος της πρώτης περίοδου δεσμεύσεων για το πρωτόκολλο του Κιώτο Έχουμε δύο προσελκύσεις, μία στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιώτο και μία στα πλαίσια της συμβάσεως. Θα έπρεπε να πετύχουμε γενική συμφωνία, θα ήταν καλύτερο για την Ευρώπη παρά να συνεχίσουμε με τη δεύτερη περίοδο υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιέτο, αλλά η κατάσταση κατάσταση η διεθνής στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία δεν διευκολύνει τα πράγματα. Στο Κανκούν απροσδόκητα καταφέραμε να προχωρήσουμε σε βασικούς τομείς που δεν περιμέναμε τότε. Όπως τη σχέση με αναπτυσσόμενες χώρες, χρηματοδότηση, μεταφορά τεχνογνωσίας, Αναμένεται ότι δεν θα πετύχουμε πλήρη συμφωνία στο Ντέρμπαν, αλλά στο Ρίο το 2012. Άρα, κατά την άποψή σας, ποια στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε να ετοιμαστούμε το ώστε στο Ρίο το 2012 τελικά να καταλήξουμε σε μια επιτυχή συμφωνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία στην οποία συμβάλατε επί της μεγάλης αυτής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ασκήθηκε από τη χώρα σας στην Ουγγαρία. Καταρχάς, έχω αυτή την ε, περιέργεια όσον αφορά την ομάδα του Βίζεγκραντ. Αναφερθήκατε στην ε, Στρόικα με την Ισπανία και το Βέλγιο, αλλά στην ομάδα του Βίζεγκραντ όπου ανήκετε έχετε κάποια πολιτική προσέγγιση, διότι επί τριών, τριών τέτοιων συνεργασιών είχαμε την Γαλλία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία πιο πριν και στην επόμενη Δανία, Κύπρος και Πολωνία. Άρα τρεις χώρες του Βίζεγκραντ θα δημιουργήσουν αυτές τις τρόικες. Ε, πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα έχει κάποια επιρροή ή όχι όσον αφορά τα ενεργειακά. Μία Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας. Αυτή η ιδέα δείχνει ότι αποκλείουν οι απόψεις όσον αφορά την εκτίμηση των πηγών ε, ενέργειας. Οι πηγές ενέργειας είναι στην αρμοδιότητα των κατών μελών. Προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσταθεμένη αξία που κομίσατε το εξάμεινο, μπορεί να μα πείτε στο μέλλον θα έχουμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέργεια, θα έχουμε κάποτε Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέργεια. Μετά, Ποια προστιθέμενη αξία πετύχατε στο εξάμεινο όσον αφορά τις υποδομές. Έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν, δεν ξέρω ποιος είναι διοκτήτης τίνος, γίνεται ένας χαμός όσον αφορά τις υποδομές. Μήπως κάποια μέρα θα πρέπει να έχουμε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που να είναι ιδιοκτήτρες των υποδομών, διότι η σωστή διαχείριση των υποδομών, κατά την άποψή μου, θα ήταν στοιχείο ανταγωνιστικότητας της υπήρου μας, κυρίως για την ηλεκτρική ενέργεια και για το φυσικό αέριο. Σα äh, Σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Κόβατς για να απαντήσει. papírjaimat azért σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω συγχαίροντας την Επιτροπή σας για τη συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή σας και την ε, Ουγγρική Προεδρία. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία αυτή και χάρη στη δική σας ε, συμβολή ξέρουμε ακριβώς ποια σημεία θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητές μας, ε, σε ποια σημεία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Θα ήθελα να ε, σας ευχηθώ να έχετε την ίδια στενή συνεργασία και με την Πολωνική Προεδρία και επιτρέψτε μου να ε, προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Ε, Κύριο Γκιούρκ, καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την Προεδρία μας με τρόπο ώστε να είμαστε φιλικοί απέναντι στο Κοινοβούλιο. Είχαμε προσπαθήσαμε να ε, ε, είμαστε παρόντες σε συνεδριάσεις ε, της Ολομέλειας και των Επιτροπών και προσπαθήσαμε να είμαστε φιλικά να απέναντι στο Κοινοβούλιο. Τώρα βέβαια επιστρέψαμε στον ρόλο του απλού κράτους μέλους, δεν έχουμε πια την Προεδρία, θα προσπαθήσουμε όμως να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πνεύμα αυτό. Ιδιαίτερα η συνεργασία του Υπουργείου μας με την Επιτροπή σας ε, ήταν πολύ θετική εμπειρία και σας ευχαριστούμε για την βοήθειά σας και για το μέλλον ως απλό κράτος μέλος, όχι ως Προεδρία πια, ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη καλή συνεργασία. Όσον αφορά τις ερωτήσεις σας, είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κάποια θέματα κλειδιά, όπως ε, το θέμα της ενιαίας καταχώρησης. Ε, στο θέμα αυτό πράγματι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας, αυτό ήταν πολύ ευτυχές γεγονός. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Μιλάμε φυσικά για το διοξίδιο του άνθρακα και την ε, ανταλλαγή σχετικών δεδομένων. Επίση, η εναρμόνιση των κυρώσεων αποτέλεσε προτεραιότητα ε, και είναι σαφέ επίτευγμα της ε, Προεδρίας μας. Επίση, η Προεδρία ενέκνε τα ψηφίσματα τη τροπολογία του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι έτσι θα συμβάλλουμε στην καλύτερη διαφάνεια, καλύτερη υποπτία τη αγορά και αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για τους ε, νέου φορεί τη αγορά. Ελπίζουμε ότι με το σύστημα τη ενιαία καταχώρηση και με την διαφάνεια στον τομέα των κυρώσεων ε, το πετυχαίνουμε αυτό. Όσον αφορά το θέμα των ποσοστώσεων του διοξιδίου του άνθρακα και τα δεδομένα που θα διατίθενται ε, και την νέα αυτή υπηρεσία που θα αναλάβει το καθήκον αυτό, καθώς και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, Νομίζω ότι και εδώ έχουμε θετικές εξελίξεις. Δεν τα ε, ανέφερα όλα αυτά στην αρχική μου ε, παρέμβαση, διότι δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Μπορώ να σας πω όμως ότι το συζητήσαμε αυτό σε, ε, στο υψηλότερο υπουργικό επίπεδο. Στις 3 Μαρτίου είχαμε μια συνάντηση στη Λουμπλιάνα είχαμε τα εγγένεια της υπηρεσίας ε, και νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος ε, θα, ε, ο αναπληρωτής διευθυντής θα έρθει εδώ στην Επιτροπή σας για να την ενημερώσει. Είχαμε και συναντήσεις με Ούγγρους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό. Όλα αυτά λοιπόν έχουν κυλήσει πολύ ομαλά. Κυρία Πολάσκα Ποπίνσκα, να απαντήσω στην ερώτησή σας. Πάντα είναι δύσκολο Καταλαβαίνετε, ένας πατέρας έχει δύο παιδιά, για ποιον είναι πιο περήφανος. Ε, είναι πολύ δύσκολο. Ε, το ανέφερα αυτό και στην αρχική μου παρέμβαση. Νομίζω ότι όλες, ε, όλα τα επιτέγματά μας ήταν σημαντικά. Να πρέπει όμως να τονίσω ένα μόνο, τότε νομίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία βρέθηκε σε πολύ ιδιαίτερη θέση, διότι στην αρχή της χρονιάς αναλάβαμε την Προεδρία για έξι μήνες και είχαμε πολύ σημαντικά θέματα στρατηγικά θέματα. Είχαμε την ενέργεια, την στρατηγική του 2020, την ε, υποδομή στον χώρο της ενέργειας. Είχαμε μια σειρά σημαντικών εγγράφων και το γεγονός ότι πετύχαμε, πετύχαμε πρόοδο ε, στα θέματα αυτά νομίζω ότι μάλλον ε, ε, είναι το θέμα για το οποίο είμαστε περισσότεροι περήφανοι. Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις στο τομέα της ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός άνευ προηγουμένου και μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό πολύ θετική εξέλιξη και για το Συμβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Το γεγονός δηλαδή ότι τόσο υψηλό επίπεδο ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά. Είναι, αυτό υπόσχεται πολλά ε, για το μέλλον. Έχουμε το 2014, το 2015, ε, την ενεργειακή αγορά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλουμε να δώσουμε τέλος στην απομόνωση ε, όσον αφορά την ε, ενέργεια. Ε, Χθε είχαμε τα τραϊκά αυτά γεγονότα στην Κύπρο, τα οποία νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι απομονωμένο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι χρειαζόμαστε αλληλεγγύη και κοινή υποδομή και γι' αυτό θεωρήσαμε τόσο σημαντικό το θέμα αυτό για την Προεδρία μας. Όσον αφορά την Πολωνική Προεδρία, τι θα προτείναμε στην Πολωνική Προεδρία. Θα ήθελα να επανέλθω σε μία παρατήρηση του Προέδρου. Η Ουγγρική Προεδρία βρέθηκε σε πολύ ιδιαίτερη θέση Αφενός διότι ήμασταν μέρος ενός πολύ επιτυχημένου τρίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου τρίο αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ήτανε είχαμε λοιπόν αυτό το προνόμιο και επίσης ε, γνωρίζαμε ότι το 2011 θα είναι ε, έτος της Κεντρικής Ευρώπης. Είχαμε τη δική μας Προεδρία, τώρα θα ακολουθήσει η Πολωνική Προεδρία και νομίζω ότι αυτό από μόνο του ε, είναι πολύ ιδιαίτερο και η συνεργασία έχει διεξαχθεί πολύ ομαλά. Για παράδειγμα, είχαμε Ήδη συζητήσει ε, με τον ε, ε, Πολωνό Υφυπουργό, η με τον Πολωνό Υπουργό. Ήταν λοιπόν πολύ καλέ οι σχέσει ανάμεσα στην Ουγγρική και την Πολωνική Προεδρία. Και επίση έχει γίνει ομαλή μετάβαση όλων των φακέλων αυτών και στι ανακοινώσει μα για την ενέργεια. Έχουμε συμβάλει και οι δύο Προεδρίες, και η Πολωνική και η Ουγγρική Προεδρία σημαντικά. Επίσης, Ε, σήμερα θα μιλήσει και ο Πολωνός Υπουργό για πολύ σημαντικά θέματα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, διότι δεν νομίζω ότι εμείς ε, πρέπει να συμβουλεύσουμε την ε, Πολωνική Προεδρία. Νομίζω ότι είναι προνόμιο τη Πολωνική Προεδρία να σκεφτεί η ίδια τι θα κάνει το επόμενο εξάμεινο. Η Πολωνική Προεδρία τώρα βρίσκεται στο φω τη Δημοσιότητα. Εκείνοι λοιπόν θα αποφασίσουν. Εκείνη αποκλειστικά δική τη απόφαση να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα θεωρήσει ότι είναι απαραίτητα. Να προχωρήσω στην ερώτηση τη κυρία Επιτρέψτε μου κυρία Τικάο να πω το εξής. Ε, το θέμα του Ναμπούκο είναι αλήθεια ότι φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση στο έργο αυτό. Σε τι βαθμό η Ουγγρική Προεδρία ήταν υπεύθυνη γι' αυτό, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω όμως ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο. Ε, βρέθηκα εκεί και ο Επίτροπος και ο Υπουργός ε, είχαμε την ε, ευκαιρία να συζητήσουμε με τις χώρες που συμμετέχουν στο Ναπούκο στην Τουρκία και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας είχε προσκαλέσει όλες τις χώρες που συμμετέχουν και τις υπηρεσίες ενέργειας Όλοι αυτοί λοιπόν ε, συναντηθήκαμε για να υπογράψουμε ε, μια συμφωνία PSA όπως λέγεται, μια συμφωνία υποστήριξη του έργου και χάρη σε αυτήν την ε, νέα συμφωνία μπορούμε να συμφωνήσουμε σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, είδαμε κάποια πρόοδο συγκεντρωθήκαμε και νομίζω ότι έτσι προωθήσαμε σημαντικά το έργο. Είμαι βέβαιος ότι και η δική σας ε, Επιτροπή εξετάζει θέματα υποδομής ε, φυσικού αερίου, διότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ο Ναμπούκο και ο Νότιος ε, Διάδρομος είναι πολύ σημαντικά έργα. Και επιτρέψτε μου, κυρία να κάνω άλλη μια παρατήρηση. Πέρα από τον αγωγό Ναμπούκο, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και για τον Βόρειο Διάδρομο, που είναι επίσης σημαντικός. Η ομάδα Visegrad 4, των τεσσάρων του Visegrad που αναφέρθηκε και από κάποιον άλλον, ε, είναι πολύ σημαντική και ε, για το σύνολο της Ευρώπης. Ε, δεν θέλαμε όμως να το αναφέρουμε αυτό ως επίτευγμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Είμαι σίγουρος όμως ότι γνωρίζετε ότι ο κύριος Μπαρόσο προσκλήθηκε σε συνάντηση με τους τέσσερις του Βίσοκρατ. Είχαμε τη Ρουμανία, την Βουλγαρία που ήταν επίσης ε, παρούσες οι χώρες αυτές ε, και συμμετείχαν σε μια ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου για να εξεταστεί η δημιουργία του αγωγού αυτού στο μέλλον. Και ε, το σημείο επαφή στην Ουγγαρία για το θέμα αυτό είμαι εγώ και γνωρίζω ότι πολλά έχουν γίνει από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες πριν από ένα χρόνο το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Ελπίζουμε ότι θα γίνει μια δεύτερη άτυπη συνάντηση και ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχουμε ένα σχέδιο δράσης για να εξετάσουμε το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και το ε, ηλεκτρικό ρεύμα. Να εξετάσουμε δηλαδή μαζί τους τρεις αυτούς τομείς ε, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε σχέδια ανάπτυξης μέχρι τότε, τα οποία θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στο μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό και για την ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού της ενέργειας και είναι και σημαντικό για την ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι ε, πολύ σημαντικό το έργο αυτό και ελπίζω ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Αυτό απαντά εν μέρη και σε άλλη ερώτηση ε, σχετικά με τον ε, συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στην ερώτηση αυτή όσον αφορά τις ανάγκες επενδύσεων. Παρακολουθήσαμε στενά τις εργασίες της Επιτροπής, ιδιαίτερα του κυρίου Έτινγκερ, και παρακολουθήσαμε στενά και τις εξελίξεις ε, γενικά. Θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει όσον αφορά το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις και θα πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες. Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε σχετικά με τις προτεραιότητες. Φυσικά δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ε, ε, επενδυτικές ανάγκες ε, με χρήματα των φορολογουμένων ή με χρήματα μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μόνο από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να συμμετάσχει. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος το ανέφερε αυτό. Έχουμε κάποιους σημαντικούς στόχους και θα πρέπει μεγάλες ενεργειακές εταιρείες Ευρώπης να συμμετάσχουν και εκείνες. Κυρία Καρβάγιο, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας η Επιτροπή Περιβάλλοντος πράγματι δεν είδε παρουσίαση της Προεδρίας. Ε, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές οι παρουσιάσεις αυτές. Είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχία σε κάποια προγράμματα και πιστεύουμε και στην πίεση που μπορεί να ασκήσει η Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε διεθνεί διαπραγματεύσει όσον αφορά τον Τέρμπαν. Έχουμε την Κίνα, έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε, έχουμε την ε, Ρωσία. Ξέρουμε ότι οι χώρε αυτέ αντιπροσωπεύουν κάποιε θέσει οι οποίε ε, δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τι δικέ μα ε, και που μπορεί να είναι επικίνδυνε. Γι' αυτό η Ένωση θα πρέπει να είναι ενωμένη απέναντι στι χωρε αυτε Στο παρελθόν, η ε, Ουγγρική Προεδρία προσπάθησε να συνδυάσει τις διάφορες απόψεις. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Νομίζω όμω ότι είχαμε κάποια επιτυχία στον τομέα αυτό και μιλάμε για δύο πράγματα. Μιλάμε για τις εσωτερικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κοιτάξτε τι έγινε στις 20 Ιουνίου. Σχεδόν πετύχαμε συμφωνία. 26 κράτη-μέλη συμφώνησαν. 26. Μόνο ένα κράτος μέλος δεν συμφώνησε. Τελικά βέβαια συμπέραψαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ε, κάποια επίμαχα σημεία. Και εμεί ω Ουγγρική Προεδρία αποτελέσαμε, ε, ε, αντιμετωπίσαμε ε, σημαντική πρόκληση στο θέμα αυτό και νομίζουμε ότι και για την Πολωνική Προεδρία ισχύει το ίδιο. Ε, τέλος, να απαντήσω στον κύριο ότι μιλήσατε για τις τρεις τρόικες. Εμείς ήμασταν το πρώτο τρίο αυτού του τύπου, τώρα ξεκινάει το δεύτερο τρίο, η δεύτερη τρόικα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποτελέσουμε παράδειγμα ή υπόδειγμα για την Πολωνική Προεδρία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, ήταν όμω ε, μεταβατική διαδικασία αυτή, από ό,τι κατάλαβα και η συνεργασία για την Πολωνία ήταν πολύ καλή. Ε, εμείς συμμετείχαμε σε τρίο με τις προηγούμενες δύο προεδρίες, ενώ η Πολωνία θα συμμετάσχει σε τρίο με τις επόμενες δύο. Ε, βλέπουμε όμως ε, τι δουλειά κάνει η Πολωνία με θέματα που ε, θα μας ενδιαφέρουν στο μέλλον. Επίσης, όσον αφορά την απόδοση της ενέργειας, το άφησα αυτό για το τέλος, διότι θα ήθελα να το αναπτύξω λίγο περισσότερο και έτσι θα κλείσω τι απαντήσει μου, διότι δεν θέλω να μακρηγορήσω το κράτησα όμως αυτό για το τέλος. Όσον αφορά την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας για το 2020, ε, Έχουμε στόχο 10%. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Κομισιόν, αντί για 20%. Και στο και πρόσφατα η Κομισιόν θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κάνει κάποια διόρθωση. Μετά από αυτό, θα έχουμε το σχέδιο απόδοσης της ενέργειας και, και αναθεώρηση του σχεδίου αυτού μετά από κάποια χρόνια και αυτή ε, η αναθεώρηση θα είναι ευκαιρία να εξετάσουμε τη στρατηγική του 2020, να εξετάσουμε τους στόχους μας, να εξετάσουμε τα εθνικά μας προγράμματα για να δούμε σε τι βαθμό είχαμε επιτυχία τελικά και τότε θα δούμε εάν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε του εθνικού στόχου. Η Κομισιόν μπορεί να υποβάλει, μπορεί και να μην υποβάλει ε, ε, νέε προτάσει, αλλά αυτό θα γίνει τότε κατά τη διάρκεια τη αναθεώρησης. Επίση, έχουμε τη θέση του Συμβουλίου και ξέρω ότι στι 22 Ιουνίου νομίζω ότι ήταν η Κομισιόν υπέβαλε έγγραφο το οποίο εξέταζε και αυτή την πτυχή και εξέταζε και άλλα θέματα τα οποία ε, μπορεί να μα ενδιαφέρουν στο μέλλον. Πάντως αυτό δεν είναι θέμα για μας που μα αφορά εμά, αφορά την Πολωνική Προεδρία ε, και τους ε, νέους αρμόδιους υπουργούς. Όσον αφορά την απόδοση της ενέργειας, ε, θα ήθελα να πω... Να κάνω μια γενική παρατήρηση. Ο δημόσιο τομέα θα πρέπει να θέσει το καλό παράδειγμα. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να Έχουμε ένα ενιαίο σημείο αναφορά. Ε, αυτό ισχύει και για την Ουγγρική κυβέρνηση. Νομίζω ε, ότι αυτό ισχύει και για όλε τι χώρε και αυτό ισχύει όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, για τι εθνικέ πρωτοβουλίε. Ε, νομίζω ότι σημαντικό είναι να το δούμε αυτό όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Και ό,τι προβλήματα ανακύψουν θα πρέπει να τα εξαλείψουμε. Και μιλάμε για τα δίκτυα, μιλάμε για την υποδομή. Θέλουμε να υπάρχουν καλά κίνητρα για τις επενδύσεις. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις και θέλουμε οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές να ενδιαφερθούν. Και φυσικά και οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς οι οποίοι μπορούν να εμπλακούν στα θέματα αυτά. Επιπλέον <clears throat> πρέπει να εμπλακούν και άλλοι παίκτες μέσα σε εισαγωγικά για να καλύψουμε όλους τους ε, ενδιαφέροντες τομείς. Τα περαιτέρω εργαλεία τώρα, τα προγράμματα αποδοτικότητα ενέργεια σε εθνικό επίπεδο στην Ουγγαρία, ήδη επεξεργαζόμαστε ένα εθνικό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση, αυτό μπορώ να σα το πω ήδη. Ε, βρίσκεται σε επίπεδο τώρα συνδιαλλαγής ε, με την κυβέρνηση αυτή η διαδικασία. Πρέπει επίσης να καταγράψουμε πιστεύω όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και να δούμε για το δρόμο το μελλοντικό. Θέλουμε να είμαστε σαφής, αποτελεσματική και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ε, αποδοτικότητα της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του βιομηχανικού τομέα, πιστεύουμε ότι οι βιομηχανίες μπορούν να έχουν πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας, ιδίω χρησιμοποιώντας το σύστημα εκπομπής εκπομπών των αρίων θερμοκηπίου. Χρειαζόμαστε επίσης ευφιέστερα ε, δίκτυα και ενεργειακά δίκτυα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, ώστε ως πολίτες και καταναλωτές να μπορούν και αυτοί να προσαρμοστούν στους νέους ενεργειακούς στόχους και να μπορέσουν να συμβάλλουν στην επιτευξή τους. Τελευταίο αλλά όχι ίστατο είναι και το θέμα του δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι απαραίτητο να υπάρξει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι πρόσφοροι στον καλύτερο δυνατό βαθμό, στον πιο αποδοτικό δυνατό βαθμό και ιδίω θα πρέπει να εντοπίσουμε τις περιοχές όπου μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες εξοικονομήσεις και μεγαλύτερη επίτευξη αποδοτικότητα συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι απήντησα σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Κόβατς για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να μεταδώσετε και στους συναδέλφους σας της Ουγγρικής Κυβέρνησης της τη βαθιά μας ευχαριστία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ καρποφόρα η συνεργασία μας παρά το γεγονός ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολα και πολύπλοκα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ναι, ίσως βιάστηκα λιγάκι. Στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης θα κάνω μια ανακοίνωση προηγουμένως Όπως σας είπα, στη γραμματεία υπάρχει συνεχής ροή, έρχονται, φεύγουν μέλη της γραμματείας συνέχεια μία αέναη αλλαγή, αλλά τώρα έχουμε δύο μέλη της γραμματείας τα οποία ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παρόντες. Η κυρία Σιλεγκόμες και η Ελένη Σαρπαντιέ. Και οι δύο ήταν για πολλά χρόνια στη γραμματεία της Επιτροπής μας έχουν υπηρετήσει σε διάφορα πόστα στη γραμματεία μας. Πάντα μπορούσαμε να τις εμπιστευόμαστε και να βασιζόμαστε σε αυτές. Έχουν δώσει πάρα πολλή ενέργεια στις εργασίες της Επιτροπής μας και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να πούμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε μαζί τους και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Thank you very much. All the best. Ωραία. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Πρόκειται για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών το 2012. Τόσες πολλές διασκέψεις έχουμε, μια παραπάνω. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω τώρα για το θέμα αυτό. Πρόκειται στην επόμενη Ολομέλεια να έχουμε μια συζήτηση για την διάσκεψη της, Ευρωπα... της ε, Παγκόσμιας ε, Υπηρεσίας ε, Τηλεπικοινωνιών για τα θέματα των ραδιοεπικοινωνιών και έχουμε συμφωνήσει με τους συντονιστές να θέσουμε ένα προφορικό ερώτημα στην Κομισιόν με συζήτηση και μετά να υπάρξει ένα ψήφισμα το οποίο βάσει του άρθρου 115 θα κατατεθεί από την Επιτροπή μας για τη λήξη της συζήτησης. Ο στόχος μας είναι τώρα να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλάει με ενία φωνή στις πολυμερείς διασκέψεις και επίσης ότι θα υπάρξει σεβασμός των αρχών της Ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισαβόνας και επίσης ότι θα παραμείνουμε πιστοί στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ε, συχνότητες και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν επαρκή τμήματα του φάσματος για τις ραδιοεπικοινωνίες, όπως τόντζε και ο κύριος Χόκμαρκ ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Χόκμαρκ, όπω είπα προηγουμένως, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Δυστυχώ δεν έχει έρθει ακόμα. Έχει καθυστερήσει. Έχουμε εδώ πέρα 26 τροπολογίε και έχουμε συμφωνήσει σε ένα κείμενο το οποίο αύριο μπορεί να περάσει στην ε, ψηφοφορία. Και εάν συμφωνείτε μπορούμε και τις 26 τροπολογίε να τι ψηφίσουμε ομού. Αν λοιπόν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση, μέχρι αύριο μπορούμε να επιταχύνουμε την ψηφοφορία, εάν συμφωνείτε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες μαζί. Τώρα δεν υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω, αλλά κυρία Τσικάου νομίζω ότι ήθελα να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τώρα κάποια παρατήρηση στην ε, πρότασή σας, απλώς θέλω να προσθέσω κάτι. Σε σχέση με αυτή την ε, διάσκεψη, δεν ξέρω αν θέλετε να το κάνω τώρα ή αργότερα. Ναι, εντάξει, μπορώ να μιλήσω τώρα λοιπόν για τη συνδιάσκεψη αυτή. Η συνδιάσκεψη αυτή για τις ραδιοεπικοινωνίες έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι εδώ διακυβεύεται το θέμα του φάσματος ε, ραδιοσυχνοτήτων και της κατανομής τους. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι ανεπαρκές αυτό το φάσμα το οποίο είναι διαθέσιμο και γι' αυτό μιλάμε για ένα σπάνιο πόρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έχει ζητήσει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και μια μεγαλύτερη εναρμόνιση στα θέματα των αδειοσυγνωτήτων για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα αυτό το τμήμα του φάσματος το οποίο διαθέσουμε. Και έχουμε διατυπώσει και μία σειρά συμπερασμάτων σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα ραδιοσυγνωτήτων για να υπάρξει ακριβώς αυτή η καλύτερη εκμετάλλευση αυτών των πόρων που είναι διαθέσιμοι, υπομορφή ραδιοσυγνωτήτων. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε περαιτέρω και για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα για το να μπορέσει, λαμβάνοντας πάντα τις αρμοδιότητες των καθών μελών και την επικουρικότητα, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό για την κατανομή των ε, συχνοτήτων του ραδιοφάσματος. Πιστεύω λοιπόν ότι στη διάσκεψη αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε και για τις παρεμβολές οι οποίες μπορούν να προκύψουν μεταξύ διαφορετικών μορφών επικοινωνιών, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές μεταξύ περιοχών μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδιαίτερα μεταξύ σε μεθοριακέ περιοχές μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της χρήσης των κινητών τηλεφώνων. Το ψήφισμά μας λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβει και κάποια στοιχεία της πολιτικής διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι εδώ στο πρόγραμμα, στο σχέδιο Γαλιλαίος και το GNSS επίσης το παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας και όπως είπα προηγουμένως η προτεραιότητά μας είναι καταρχήν η κατανομή του ραδιοφάσματος αλλά δεύτερον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα των παρεμβολών στο ραδιοφάσμα που μπορούν να προκύψουν. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Α, ο κύριος Χαρκμακ θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, θα τα πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ένα τουριστικό λεωφορείο ε, ήταν που με έφερε έξω από αυτό το κτίριο και χρειάστηκε και κάποιο χρόνο για να ανέβω τα αλκυστήρα. Για την πρόταση ψηφίσματο να πω κάποια πράγματα για το κείμενο. Ήταν αρκετά εύκολο να συμφωνήσουμε. Το κείμενο την χάνει ευρεία υποστηρίξεω από όλε τις πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια και πρέπει να υπογραμμιστεί, διότι κάποια από αυτά τα θέματα είναι μάλλον επίμαχα. Και δείχνει το αποτέλεσμα ότι τελευταίου μήνες συζητήσαμε αρκετά καλά τι ανάγκε των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των φασμάτων, των δυσοκνοτήτων. Όσον αφορά τη διάσκεψη για τα θέματα αυτά, το 2012 έκανε θετική σημασία στη διάσκεψη. Υπάρχουν πιεστικέ ανάγκε. Πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα των συχνοτήτων και η απόφαση που θα ληφθεί στην επόμενη διάσκεψη για τις συχνότητες του 2015 θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμα εργασιών και το 2012, στην ημερήσια διάταξη του 2012. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των, του σφάσματος των συχνοτήτων. Είχαμε εξετάσει το θέμα και θετήσαμε ένα κείμενο πριν από μερικούς μήνες στο Κοινοβούλιο. υπήρξε ευρεία συνεννόηση όσον αφορά το κείμενο του ψηφίσματο. Έγιναν αποδεκτέ διάφορε απόψει και διάφορε οπτικέ γωνίε των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Άρα δεν χρειάζεται να το πολύ κουβεντιάσουμε. Σημειώνουμε ότι ήταν εύκολο το έργο μας. Και ευχαριστώ γι' αυτό όλους τους εκπροσώπους των άλλων ομάδων επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, να προσθέσω κάτι κυρία Πρόεδρε. Μία σκέψη. Δεν αναφέρεται στο ψήφισμα. Ίσως είναι τροφή προσκέψη στο μέλλον. Το φάσμα. Οι τηλεπικοινωνίες. Είναι τομεί που αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα στη σύγχρονη κοινωνία. Και είναι παράξενο το ότι σε αυτό το τομέα η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλη Κάθε τρία-τέσσερα χρόνια γίνεται αυτή η διάσκεψη για τι ραδιοσυχνότητε. Και όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Ακολουθούμε παράδοση δεκαετία του 20 του περασμένου αιώνα. Στο μέλλον θα πρέπει να το σκεφτούμε πώ θα πρέπει να κινούμαστε όσον αφορά αυτέ τι αποφάσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά αυτό το ψήφισμα, κάτι για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν έξυπνο αυτό το οποίο αναφέρετε και η διαδικασία είναι πάρα πολύ σαφή. Ψηφίζουμε όπω είπα αύριο. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, το σημείο 6. Και θέλω να χαιρετήσω τους καλεσμένους μας και συγκεκριμένα τον κύριο Ποτόσνικ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Acer. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε όποτε είσαστε έτοιμος κύριε Ποτόσνικ, όταν έρθετε εδώ. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι σήμερα καλωσορίζω μια σειρά προσκεκλημένων πέρα από τον κύριο Ποτότσνικ, που είναι Διευθυντής του Οργανισμού Συνεργασίας ε, των Ρυθμιστικών Αρχών ε, Ενέργεια. Ε, καλωσορίζω και τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών, που έχουν έρθει εδώ σήμερα. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποτότσνικ. Κατόπιν θα ακολουθήσει η συζήτηση. Μόνο να φροντίσουμε να προλάβουμε και τα άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να ε, έχετε κατά νου σας και την ώρα. Κύριε Ποτόσνικ, ε, σας καλωσορίζω. Μπορείτε να ξεκινήσετε αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κρυμμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Είχα παρόμοια δυνατότητα εδώ και ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2010, μετά που ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν διευθυντή υπηρεσία για τη συνεργασία όσον αφορά τον φορέα των εθνιστικών τομέα τη ενέργεια και τότε συζητούσαμε τι προσδοκίε σα και τα σχέδιά μου. Και χαίρομαι που λέω ότι σήμερα είμαι σε θέση να παρουσιάσω κάποια αρχικά επιτέγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ο φορέα μέχρι τώρα. Μαζί μου Έχω τον Λόρδο Μόγ, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Φορέων της Υπηρεσίας και πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Φορέων Ρύθμισης και τον Βότερ Μπόλτς, που είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος του CR. E λοιπόν, αυτό που θα κάνω θα είναι να διατρέξω τις εξελίξεις στο, στην υπηρεσία μας πώς ε, ολοκληρώνουμε, πώς εφαρμόζουμε το πρόγραμμα εργασιών μας για φέτος και πώς παρουσιάζουμε το πρόγραμμα εργασιών για τον επόμενο χρόνο. Πολύ πρόσφατα υιοθετήθηκε το πρόγραμμα για τον χρόνο και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από την προηγούμενη παρουσίασή μου εδώ ήμασταν σε επαφή. Δημιουργήσατε μια ομάδα επαφής ASA και ήμασταν σε επαφή με αυτή την ομάδα επαφών, επαφής μάλλον το Δεκέμβριο ε, έχουμε διανύμει, είχαμε διανύμει τότε και μια έκθεση προόδου και η παρουσίασή μου στο φόρουμ της Φλωρεντίας ε, διενεμήθη επίσης τα μέλη της ομάδας επαφής. Ήμασταν σε επαφή αλλά είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι παρόν εδώ σήμερα. Λοιπόν, αν δούμε λοιπόν τι συνέβη μέχρι τώρα, ανέλαβα τη θέση μου στις Βρυξέλλες, τα καθήκοντά μου μέσα Σεπτεμβρίου πέρσι και τον Οκτώβριο η ομάδα άρχισε να δημιουργείται αρκετά γρήγορα από την ανάληψη των καθηκόντων μας. Στις 26 Νοεμβρίου μπορέσαμε να υπογράψουμε τη συμφωνία για την έδρα μεταξύ τη υπηρεσία τη κυβερνήσεω της Σλοβενίας και πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προ τη σλοβενική κυβέρνηση για τη στάση που ετήρησε. Ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη και κράτησε αυτή τη στάση καθ' όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων τη συμφωνία. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο και μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει και να υπογράψουμε τέλο Νευρίου. Αυτό σημαίνει ότι ε, μέχρι την 1η Δευτέρου 2011 μπορέσαμε να μετακομίσουμε, να πάμε στη Λιουμπλιάνα και λειτουργούμε στη Λουμπλιάνα έκτοτε. Όπως ήδη θα ακούσατε και από την Ουγγρική κυβέρνηση ε, αρχίσαμε να λειτουργούμε επίσημα στις 3 Μαρτίου φέτος όπως ετέθησε ισχύ και το τρίτο ενεργειακό πακέτο την ίδια στιγμή. Εγκαινιάσαμε τα γραφεία μας στη Λουμπλιάνα, βλέπετε εκεί με κόκκινο, στο κόκκινο τετράγωνο, βλέπετε τα γραφεία μας και βλέπετε και κάποιες εικόνες από την εκδήλωση οπότε λειτουργούμε από τον Μάρτιο στην Λουμπλιάνα και εκεί εδρεύει η ομάδα μας. Λοιπόν, όσον αφορά τις προσλήψεις, ξεκινήσαμε τις προσλήψεις πέρσι. Άρχισαν οι προσλήψεις και πριν μπω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησαν οι προσλήψεις και πρέπει να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια και άλλες γενικές διευθύνσεις για την υποστήριξη που μας παρίσχουν κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας το προσωπικό μας είναι 52 άτομα, εγώ συν 51 άλλα μέλη, 10 από αυτά ε, θα έρθουν ή έρχονται σαν αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Σε αυτή τη χρονική περίοδο έχουμε ήδη 23 άτομα που εργάζονται στα γραφεία μας στη Λουμπλιάνα και ένα στο γραφείο επαφής στις Βρυξέλλες που άνοιξε πριν από ένα δίμηνο περίπου. Έχουμε άλλους 8, άλλα 8 μέλη που ήδη έχουν διοριστεί και ήδη έχουν ε, μία ημερομηνία που θα ξεκινήσουν να δουλεύουν από τώρα με τον Οκτώβριο και έχουμε ήδη δρομολογήσει διαδικασία προσλήψεων για άλλες 16 θέσεις αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου με ενδεχόμενη εξαίρεση μίας θέσης. Μέχρι το τέλος του χρόνου ε, θα έχουμε 51 ή συνολικά 52 θέσεις καλυμμένες και το προσωπικό που θα εργάζεται στη Λουμπλιάνα. Τώρα, οι εθνικότητες δεν ήταν κριτήριο η επικότητα για την επιλογή του προσωπικού, δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, όμως σαν αποτέλεσμα των διαδικασιών επιλογής μέχρι τώρα, έχουμε αρκετά ποικίλο φάσμα όσον αφορά τις υπηκότητες του προσωπικού και χαίρομαι που λέω ότι είναι μια πτυχή αυτή που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τη δουλειά της υπηρεσίας. Παρόλο λοιπόν που δεν ήταν στόχος αυτός καθεαυτός. Είμαστε αρκετά τυχεροί και σήμερα έχουμε αρκετά ευρύ φάσμα ε, Ευρωπαίων από διάφορες χώρες που εργάζονται για τον οργανισμό μας. Θα ήθελα να στραφώ τώρα προς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε το πρόγραμμα εργασιών για φέτος. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, ε, έλαβαν χώρα αρκετές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του προγράμματος εργασιών του 2011, γνωμοδοτήσεις όσον αφορά τα καταστατικά και κατάλογο εσωτερικός κανονισμός, μέλη κλπ. για το enso e και το ΕΝΤΣΟΚ, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά σαν νέα θεσμικ... νέοι θεσμικοί φορείς, κατευθυντήριες γραμμές, προσανατολισμοί, είναι διάφορα έγγραφα που περιέχουν τα κριτήρια και τις διάφορες αρχές που πρέπει να εφαρμοστούν και είχαμε οκτώ κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο πρόγραμμα εργασιών για φέτος και πρέπει να ολοκληρωθούν. Έχουμε επίσης ε, γνωμοδοτήσεις και συστάσεις όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών των δύο έντσο και για το δεκαετές πρόγραμμα αναπτύξεως των δικτύων. Έχουμε εντολή ε, για να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο Αντιστάθμισης μεταξύ των έντσο λειτουργεί παρόπου αφαιρέθηκε αυτό το στοιχείο αργότερα από το πρόγραμμά μας μέσω νέου κανονισμού, ο οποίος μας δίνει και άλλες συμπληρωματικέ ευθύνε, αλλά στη διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και μετά έχουμε ευθύνε όσον αφορά τον έλεγχο της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και έχουμε και ευθύνε όσον αφορά την παρακολούθηση της περιφερειακής συνεργασίας και αυτές οι δύο πτυχές είναι κάτι που προετοιμάζουμε για να ξεκινήσουμε την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας από του χρόνου και ήδη υπήρξαμε αρκετά δραστήριοι όσον αφορά τις περιφερειακές ε, πρωτοβουλίες. Τώρα όσον αφορά το τι πετύχαμε μέχρι τώρα βλέπετε γραφική παρουσίαση, ε, εικονική παρουσίαση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι απομένει για το υπόλοιπο του έτους. Εστιαζόμεθα επί των καθετηρίων γραμμών που αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα που είναι και το σημαντικότερο στοιχείο το σημαντικότερο αποτέλεσμα του οργανισμού μας για φέτος και χάρη θα έλεγα στην συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ΕΡΓΕΡ και την CR μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τις δημόσιες διαβουλεύσεις επί δύο ε, σχεδίων προσανατολισμών την ίδια ημέρα όπως ε, τις 3 Μαρτίου που ξεκίνησε και επίσημα τις εργασίες της οργανισμός μας. Η δουλειά συνεχίζεται ομαλά όσον αφορά αυτούς τους προσανατολισμούς και μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές Αυγούστου θα μπορέσουμε ήδη να εκδώσουμε τρεις προσανατολισμούς για την ώρα. Έχουμε δώσει ήδη την γνωμοδότησή μας όσον αφορά το καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό και κατάλογο μελών των δύο έντσο, ούτω ώστε έχουν ό,τι χρειάζονται τόσο ώστε να λειτουργούν σωστά στα πλαίσια του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Υπάρχουν άλλες κατευθυντήριες γραμμές ρυθμιστικές στο πρόγραμμα εργασιών για φέτος, όπου για την ώρα τα επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία και θα γίνει και δημόσια διαβούλευση σχετικά αργότερα το τρέχον έτος. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα για του χρόνου, Ένα μέρος αυτού θα αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων του ενεστώτος έτους και όπως γνωρίζετε από τη στιγμή που θα εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραμμές πλαίσιο και θα υιοθετηθούν από τον οργανισμό, θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαβιβαστούν στις έντσο, οι έντσο θα δημιουργήσουν τους διάφορους κωδικούς για το δίκτυο που θα επιστρέψουν στον οργανισμό, τόσο ώστε ο οργανισμός να κάνει την αξιολόγηση και να δει κατά πόσο συμμορφώνονται αυτές τις προτάσεις με τις αρχές και τα κριτήρια των κατευθυντηρίων γραμμών πλαίσια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επεξεργασία των κατευθυντηρίων γραμμών Μία-δύο από αυτές θα αφορούν διαλειτουργικότητα, εξισορρόπηση όσον αφορά το φυσικό αέριο και θα μεταφερθούν οι προσπάθειες από φέτος τον επόμενο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε και νέα σημεία πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια τρίτων μερών, κανόνες για εμπόριο και ανταλλαγή στοιχείων και καθορισμός κανόνων για το φυσικό αέριο και θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε και το διάφορους κώδικες για τα δίκτυα και περιμένουμε να δούμε διάφορους κώδικες από την ENSO ή και ENSOC να εξετάσουμε τις προτάσεις που προταθούν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση και υιοθετηθούν μέσω της διαδικασίας ε, επιτροπολογίας. Θα εξετάσουμε επίσης, θα δώσουμε γνωμοδότηση και σύσταση όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών των δύο έντσο και το πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων, το δεκαετές πρόγραμμα φέτος θα λάβουμε πολύ σύντομα και μια πρόταση για το φυσικό αέριο και του χρόνου αναμένεται να λάβουμε την πρόταση για την ηλεκτρική ενέργεια. Παράγονται κάθε διετία αυτές οι προτάσεις και την χάνει ότι θα παραληφθούν σε ξεχωριστά έτη. Επίσης, εξετάζουμε και τον έλεγχο της δραστηριότητε της ελεγκτικές, της εσωτερικής αγοράς, της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Φέτος, όπως ανέφερα, θέλουμε να δημιουργήσουμε δείκτες και παραμέτρους για να αρχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις του χρόνου στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Αυτές είναι δραστηριότητε πριν η αδίποτε εφαρμογή της εντολής, εκτέλεση εντολής. Μία από τις άλλες στοιχείες που όλο και περισσότερο γίνεται σημαντική είναι οι περιφερειακές πρωτοβουλίες και η διάσταση αυτών με την εφαρμογή των κανόνων για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η περιφερειακή διάσταση γίνεται ξανά πολύ σημαντική και εξετάζαμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προωθήσουμε τη συνεργασία. Και τέλος η ε, εντολή που δόθηκε παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις εντός του Συμβουλίου και εντός του Κοινοβουλίου και προετοιμαζόμαστε για να εφαρμόσουμε τον κανονισμό ε, όποτε θα υιοθετηθεί Ετοιμάσαμε ήδη προπαρασκευαστικές εργασίε και θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε και σχετικέ δραστηριότητες που θα πρέπει να δρομολογήσουμε. Αυτή είναι η παρουσίαση. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προφανώς κύριε Πρόεδρε με τα χαράς και, συνάδελ... οι συνάδελφοί μου και εγώ να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Ήταν πολύ σαφή αυτά που μα είπατε. Ωστόσο υπάρχουν κάποιε ερωτήσει. Καταρχήν ο συνάδελφο Γκιόρκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Διευθυντά, για την παρουσίαση αυτή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Στο προηγούμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, μιλήσαμε για την ε, Ουγγρική Προεδρία και το τι κατάφερε. Και Επίσης αναφερθήκαμε στην ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και εκφράσαμε μια ελπίδα. Ε, τουλάχιστον εγώ το έκανα αυτό. Ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Και ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια αυτά που ελπίζουμε θα γίνουν πραγματικότητα, η ενιαία αγορά ενέργειας για την Ευρώπη. Νομίζω ότι έχετε να παίξετε ρόλο κλειδί στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να εργαστείτε με επιτυχία εάν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά ενέργειας στο μέλλον. Όσον αφορά ναι. το τελευταίο σας θέμα, το REMIT, ναι. νομίζω ότι ε, αυτό ε, θα μπορέσει να αποτελέσει ε, την αποφασιστική δοκιμή για το όλο θέμα. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ και γι' αυτό τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις για το REMIT Έχοντας αυτό λοιπόν κατά νου θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Όσον αφορά τις, ε, την, όσον αφορά την εποπτεία, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Στην καθημερινή εποπτεία, τι επιπλέον καθήκοντα προβλέπετε για το μέλλον, δηλαδή τι δεν έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα, τι πιστεύετε ότι ε, απομένει να γίνει πέρα από τα όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Και επίσης πιστεύετε ότι θα έχετε τους απαραίτητους πόρους, το απαραίτητο δυναμικό για να μπορείτε να κάνετε αποτελεσματικά τη δουλειά σας στο μέλλον. Ε, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον πόρους, αυτό είναι, αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Ε, άλλη ερώτηση που συνδέεται με την πρώτη. Είμαι βέβαιος ότι έχετε παρακολουθήσει τις νομοθετικές εξελίξεις, ότι έχετε, ότι έχετε εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής και θα έχετε δει ότι σε πολλούς τομείς έχουμε προχωρήσει πέρα από αυτά που ήλπιζε η Επιτροπή. Τώρα λοιπόν θα πρέπει οι απαιτήσει αυτέ να εισαχθούν στι ε, χώρε όπου δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σε κάποιε χώρε δεν υπήρχε ενιαία καταχώρηση. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ακούσω την ε, δική σα άποψη σχετικά με το νέο αυτό σύστημα. Πώ πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει στην πράξη. Και έχω μια τρίτη ερώτηση πάλι για το REMIT. σε αρκετά κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι Υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες ε, με χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Τι θα γίνει με αυτές στο μέλλον, για παράδειγμα πώς μπορούμε να αποφύγουμε αρνητικές συνέπειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη παρουσίαση που κάνανε για την ε, δραστηριότητά τους ενώπιον των Ευρωπαϊκών ενώπιον της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ήμουν παρόν στην έναρξη των δραστηριοτήτων του φορέα αυτού στη Λουμπλιάνα και διεπίστωσα ότι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εργασία τους και όλα πάνε καλά. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλό συντονισμό όλων των εθνικών ρυθμιστών στα θέματα ενέργειας, ώστε να συμβάλλει αυτή η συνεργασία σε μια καλύτερη ανάπτυξη της ε, αηφόρχωσης της ενέργειας στην Ευρώπη και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας και αυτό αφορά ιδιαίτερα ε, <clears throat> την συμπλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η καλύτερη συνεργασία όλων των ενεργειακών συστημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχει και ο στόχος να υπάρξει και καλύτερη χρήση των ενδικτών σε σχέση με την χρήση της ενέργειας. Ξέρετε επίσης ότι πέραν των προτάσεων που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν και οι προσπάθειες των ε, ρυθμιστών της ε, Acer που επίσης είχαν να αντιμετωπίσουν μερικές φορές τη δυσπιστία και την αντίδραση ορισμένων κρατών μελών. <clears throat> και είχαν και δυσκολίες με ορισμένες ρήτρες της Συνδίκης Λισαβόνας. Γι' αυτό η Acer χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες. Και φυσικά υπήρξαν και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πολλές φορές λαμβάνουν χώρα στις μεθοριακές περιοχές μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι έχει καταφέρει η Acer να βρει συγκεκριμένες και επιτυχείς λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι πάρα πολλά εξαρτώνται από την σωστή λειτουργία του φορέα αυτού. Χρειάζεται να προωθήσει και την φιλελευθερωποίηση προς το κοινό των καταναλωτών, να δοθούν κίνητρα στους επενδυτές και να υπάρξει μια υποστήριξη να, να προωθηθούν καλύτερες μορφές ε, λειτουργίας των δικτύων σε χώρες ιδίως όπως η δική μου, η Ρουμανία. Γιατί η Ρουμανία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πολλά προβλήματα διότι ο τρόπος με τον οποίο είχε γίνει η κατανομή των συμβάσεων δεν ήταν πάντα ο καλύτερος δυνατός στη Ρουμανία <clears throat> και δεν αποσκοπούσε μονάχα στην καλύτερη χρήση της ενέργειας. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι αγόραζαν ενέργεια και μετά τη μεταπολούσαν και είχαν σημαντικό περιθώριο κέρδους από αυτές τις ενέργειες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των τιμών και όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Και λαμβάνοντας υπόψη την ε, νέα στρατηγική της, Ευρωπαϊκής, της Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογραμμίσει ο Επίτροπος Ρούτιγκερ ότι θα πρέπει όλα τα κατημέλη να προσαρμόσουν την, ε, το κανονιστικό της πλαίσιο και τις ρυθμίσεις του στην, ε, στην, στις προδιαγραφές και στις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες χώρες λοιπόν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και θα ήθελα να ξέρω τι μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλιστεί ότι οι χώρες αυτές θα κάνουν μια ταχύτερη προσαρμογή της νομοθεσίας τους. Και πιστεύω ότι όλες οι διαδικασίες διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι συνεκτικές και διαφανείς, αλλά θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει και ευρύτερος αντίκτυπος προς την κοινή γνώμη, να υπάρξουν λοιπόν εργαστήρια και σεμινάρια μέσω των οποίων θα μπορέσει η Acer να συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πολύ λίγοι από τους ε, καταναλωτές, δηλαδή τα, τα νοικοκυριά στην Ευρώπη, που γνωρίζουν πράγματι ποια είναι τα δικαιώματά τους. Και επομένως δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους, να τα διεκδικήσουν. Κάποια μελέτη κατέδειξε ότι μόνο 12% των Ευρωπαίων καταναλωτών άλλαξαν πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών με τη φιλελευθεροποίηση. Και πρέπει λοιπόν ο καταναλωτής να πληροφορηθεί καλύτερα για τη δυνατότητα βελτίωσης της ενεργητικής απόδοσης. Εν τέλει θέλω να καταγράψω επίσης και το γεγονός ότι για μένα η Acer θα πρέπει να είναι μια πηγή μόνιμου διαλόγου και να έχει μόνιμη επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε και εμείς να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε αυτό το φορέα να επιτύχει τους στόχους τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ε, ένας αριθμός εθνικών αριθμιστών. Ελπίζω λοιπόν ότι η Acer θα μπορέσει να επιτύχει όλους τους φιλόδοξους στόχους που έχει διατυπώσει και ότι θα είναι σε θέση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων όπως προβλέπεται και στο πρόγραμμά της της 2012. Είναι η ελπίδα μου λοιπόν ότι οι δραστηριότητες του φορέα σας θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κλοντ Τσούρμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά και κύριε Υποδιευθυντή, θα ήθελα καταρχήν να ομολογήσω ότι έχω εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα με την οποία καταφέρατε να ε, δημιουργήσετε, την, να στήσετε αυτή την υπηρεσία. Επίσης το πρόγραμμα εργασίας σας για το 2011 φαίνεται επίσης να λειτουργεί ομαλά. Σα ευχαριστώ και πάλι που δημιουργήσατε ένα γραφείο επαφή στις Βρυξέλλε. Ε, ήταν ένα από τα θέματα στα οποία είχα επιμείνει, διότι νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσετε να διαδώσετε αυτά που κάνετε στη Λιουμπλιάνα και να βρίσκεστε κοντά στο κέντρο των αποφάσεων. Ε, έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχήν, η Κομισιόν στο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ήθελε να διαθέσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, ενεργειακή υποδομή. Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειαζόμαστε τόσα χρήματα, διότι για μένα είναι ε, ρυθμισμένο θέμα η ενεργειακή υποδομή. Είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ποια είναι η δική σας συμβουλή προς την Κομισιόν Εάν δώσουμε κάποιες ε, άμεσες ε, επιχορηγήσεις, ε, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια για να πει υπάρχει στρέβλωση. Εάν λοιπόν δώσουμε, εάν επιχορηγήσουμε μια υποδομή, αυτό σημαίνει ότι θα εισπράττει λιγότερα ο οικονομικός φορέας ε, διότι αλλιώς ε, θα πληρώνετε δύο φορέ, μία φορά από τον φορολογούμενο και άλλη μία φορά από τον καταναλωτή. Δεύτερον, μπορείτε παρακαλώ να ε, αναπτύξετε το θέμα αυτή της αποζημίωσης που αναφέρατε, της NTSO, διότι αυτό πώς σχετίζεται με την διασυνοριακή κατανομή των εξόδων Κάποιοι λένε ότι χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό για να γίνει ε, κατανομή διασυνοριακή των, του κόστους ε, των υποδομών. Έχετε κάτι να μου πείτε για το θέμα αυτό. Τρίτον, όσον αφορά την ε, αγορά φυσικού αερίου, πάντα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι επενδύουμε τόσα χρήματα στους αγωγούς εκτός της Ευρώπης και τόσο λίγα επενδύουμε εντός της Ευρώπης για την ροή του φυσικού αερίου από ένα μέρος στο άλλο. Τι κάνετε για να βελτιώσετε την ε, εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Τέταρτον, όσον αφορά την ε, ανταπόκριση στην ε, ζήτηση. Και Όσον αφορά τον ε, ηλεκτρισμό, ε, ε, εμποδίζουμε ουσιαστικά τις νέες επενδύσεις. Δεν έχω δει τίποτα σχετικό. Αυτό το έχετε αναβάλει για του χρόνου και τέλος. όσον αφορά τους λειτουργούς των συστημάτων διανομής. Συμφωνούμε ότι σε επίπεδο TSO χρειαζόμαστε περισσότερα, αλλά όσον αφορά τους διανομής σε όλο αυτό το παιχνίδι εξυγχρονισμού της υποδομής ε, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πού βρίσκονται αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να δώσω τώρα τον λόγο σε ένα μέλος της Επιτροπής μας που έχει γίνει αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπετε, μερικές φορές μπορεί κανείς ε, να έχει εξαιρετική ε, σταδιοδρομία όντας μέλος της Επιτροπής μας. Τζάιλ, ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευγενική αυτή εισαγωγή. Ήμουνα πρόεδρος της Επιτροπής αυτής και ήταν αυτό πολύ απαιτητικό έργο, οπότε η μόνη μου φιλοδοξία μετά ήταν να γίνω αντιπρόεδρος ε, μας είπατε να έχουμε κατά νου την ώρα ε, και κοίταζα εδώ πέρα το ρολόι και έλεγα μα, και σκέφτηκα ότι μα τόση ώρα μιλάει, μήπως ε, θα θέλατε να μηδενίσετε το ρολόι. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, ε, σημείωσα την ώρα, δεν ε, μακρηγορήσατε, αλλά θα πρέπει να είμαστε ε, δίκαιοι στα θέματα αυτά. Πρέπει να το πω αυτό ως Αντιπρόεδρος. Ε, κύριε Ποτόσνικ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι στην ε, νομοθεσία εισάγαμε τη δυνατότητα να παρουσιάζεστε εδώ στην Επιτροπή μας και να ακούτε τις απόψεις μας, να χρησιμοποιείτε την Επιτροπή μας ε, ως πλατφόρμα για θέματα που θέλετε να θίξετε και να διαδώσετε. Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ότι ε, κανένα νέο είναι καλά νέα, διότι φαίνεται να μην έχετε σημαντικά προβλήματα. Αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί όμως κάποια στιγμή να θεωρήσετε χρήσιμο να έρθετε στην Επιτροπή μας πέρα από τις επαφές σας με την Επιτροπή. Έτσι μπορείτε να διατηρείτε και την ε, ανεξαρτησία σας, την αυτονομία σας, ε, η οποία είναι πολύ σημαντική. Επίσης, με ενδιαφέρει το δεκαετές ε, πρόγραμμα ανάπτυξης. διότι η ενέργεια είναι μακροπρόθεσμη υπόθεση και αναρωτιέμαι εάν έχετε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την πρόοδο αυτών των αναπτυξιακών σχεδίων. Αναρωτιέμαι αν έχουν προκύψει νέα στοιχεία και αν πιστεύετε ότι η δεκαετία είναι κατάλληλο χρονικό διάστημα Στην σχετική οδηγία, όταν ήμουν εισηγητής, ε, εμείς ε, είχαμε την 15η ως χρονικό διάστημα, διότι θεωρούσα ότι αυτό είναι το διάστημα που απαιτείται για τη δημιουργία νέας υποδομής ε, ω ανταπόκριση στις αλλαγές στην αγορά. Έχετε λοιπόν νέα στοιχεία και ως νομοθέτες, ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε με το θέμα της ε, διανομής. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, ε, χαίρομαι που μαθαίνω ότι πήγανε πολύ καλά τα πράγματα με τη σχετική συμφωνία σχετικά με την έδρα σας, διότι είμαι μέλος του Κοινοβουλίου που ασχολείται με τις υπηρεσίες και τις ε, σχέσεις τους με τις χώρες ε, όπου εδρεύουν. Και όπως γνωρίζετε κάποιες από τις υπηρεσίες, ε, κάποιους, κάποιοι από τους οργανισμούς αυτούς βρίσκονται πολύ μακριά από τις Βρυξέλλες και θα θυμάστε ότι εμείς είχαμε προτείνει η δική σας υπηρεσία να βρίσκεται εντός των Βρυξελών. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω ρωτήσω εάν ε, έχετε περαιτέρω σχόλια όσον αφορά την ε, συμφωνία αυτή για την έδρα σας. Ε, και πέρα από αυτό θέλω να πω ότι χαίρομαι που τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Τρίτη με ερώτηση. Αφορά το ρόλο της υπηρεσίας ε, σε περίπτωση κάποιου γεγονότος σε νήμιον 1. Ε, Φυσικά είναι θέμα που ενδιαφέρει ε, αυτούς ε, που ε, χειρίζονται το σύστημα διαβίβασης. Αναρωτιέμαι τι θα κάνετε σε κάποια περίπτωση. Έχω ακούσει φήμες ότι πρόσφατα σε κάποιο κράτος μέλος είχαμε ένα τέτοιο γεγονός. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Εγώ αναφερόμουν σε ένα κράτος μέλος στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ Κλωτ, πάντως για την παρέμβασή σου. Μου θύμισε ο Κλοντ Πάντω ότι είχαμε και ένα πρόβλημα σε κράτος μέλος που έχει υποσχεθεί να, ε, να, κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια. Αλλά πάση πτώση, η ερώτησή μου είναι πώς ε, βλέπετε εσείς τον ρόλο της ε, υπηρεσίας και των νομοθετών σε μια τέτοια περίπτωση. θα πρέπει απλά να παρακολουθούμε την κατάσταση ή θα πρέπει να συμμετάσχουμε στον όλο συντονισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα σας ξαναδώσω λοιπόν τον λόγο κύριε Ποτόσνη, γιατί είδατε ότι υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα ερωτήσεων που απευθύνθηκε σε εσά. Μπορώ και εγώ να προσθέσω και ο κύριος Μόξτατ ίσως. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Μόξτατ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Τσίτσεστερ που έχει αναλάβει τη θέση αντιπροέδρου. Υπάρχουν μερικοί από εμά που είμαστε αρκετά μεγάλοι και θυμόμαστε ότι έχουμε υπηρετήσει υπό την Προεδρία του αυτή την Επιτροπή. Αξίζει τα πάντα όλες τις επιτυχίες που έχει καταφέρει. Ζήτησα το λόγο πρώτος για να πω το εξή ότι εκ μέρου πολλών συναδέλφων πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας. Δεν είναι λόγια κολακίας, Είμαστε ευγνώμονε προ την Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο σχετικά με αυτά που έκαναν για την ενέργεια τα τελευταία χρόνια. Αυτή η προσπάθεια ε, βελτίωσε πολύ την γενικότερη θέση και του οργανισμού μας, αλλά και προωθήθηκε και ο ενεργειακό τομέα με αυτέ τι προσπάθειε. Να υπογραμμίσω και κάτι άλλο, που αφορά και μια-δύο ερωτήσει που ετέθησαν. Υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών και του οργανισμού μας. Αυτό αποδεικνύεται επικοιλωτρόπως. Κατά την ενδιάμεση περίοδο που εφαρμοζόταν η νομοθεσία, οι εθνικές εθνιστικές αρχές εργάστηκαν σαν να υπήρχε ο οργανισμός. Οπότε ο, ο φόρτος εργασίας του οργανισμού αντικατοπτρίζει και τις, το έργο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν τους πόρους τους στον οργανισμό μας μέσω μιας περίπλοκης διαδικασίας. Μας βοήθησαν όσο αφορά αίθουσες, συνεδρίασεις κλπ, κτίρια και έτσι λειτουργούμε αποτελεσματικά, γιατί μα διαθέτουν χώρους εδώ και λειτουργούμε σε ελάχιστο κόστος. Αυτή η συνεργασία σημαίνει ότι υπάρχει συνεργασία και με τι εθνικέ εθνιστικέ αρχέ που εργάζονται εντό του οργανισμού, διότι εξάλλου εντό του πλαισίου μα εργάζονται εθνικέ εθνιστικέ αρχέ και μέσω τη ΣΥΑ στο εξωτερικό επίπεδο, στην πραγματική σχέση και ουχή ανταγωνιστική. Σαν πρόεδρο και των δύο φορέων, πρέπει να πω ότι δεν είδα κανένα στοιχείο και ελπίζω να μην δω ποτέ κανένα στοιχείο, λέγω, ανταγωνισμού. Ας αφήσω το πρώτο ερώτημα και ας πάω στο δεύτερο, του κυρίου Λέντσιου. Συντονισμός. Υπάρχει σαφής βελτίωση όσον αφορά το συντονισμό. Πρώτα απ' όλα γιατί συναντιόμαστε συχνά. Τουλάχιστον δύο μέρες το μήνα, καμιά φορά και συχνότερα. Και η ένταση συνεργασία, ο επίπεδο ομάδα εργασία είναι εξουσιομοιώτη. Μα υποχρεώνεται αυτή η συνάντηση. Το τρίτο πακέτο έχει αυτή την κατεύθυνση. Αλλά έχουμε και πολλέ προκλήσει στον ενεργειακό τομέα, το ξέρετε καλά. Τεράστιε προκλήσει. Υπάρχουν και άλλοι τομεί όμω όπου εργαζόμαστε ξεχωριστά από τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ. Για παραδείγματι, οι διεθνείς πτυχές, περιορισμένοι πόροι που έχει ο Αλμπέρτο στον οργανισμό, σημαίνουν ότι εμεί αριθμιστικοί φορεί πρέπει να καλύψουμε το κενό και να έχουμε καλέ σχέσει και με πολυμερείς φορείς αλλά και με χώρες μεμονωμένες όπως Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτά που συμφώνησε στο τρίτο πακέτο το Κοινοβούλιο να εφαρμοστούν και σωστά. Τι μας προβληματίζει ότι στην εφαρμογή τα κράτη-μέλη ίσως δεν πετύχουν, έχουν ανεξαρτησία η εθνική ρυθμιστική φορείς σε κάποιες χώρες και ελπίζω το Κοινοβούλιο να εξετάσει του αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιεί σωστά τα όσα έχουν ζητηθεί. Τρίτος τομέας, ακροθυγός, αύξηση αρμοδιοτήτων. Κάποια κράτη-μέλη έχουν αντίρρηση γι' αυτό. Ας αφήσουμε τα θέματα κυριαρχίας παράμερα για την ώρα. Και εφόσον ο μυστικός φορές δεν αναφέρονται στα πολιτικά θέματα, η διάσταση της συνεργασίας, το μέγεθος της συνεργασίας, μας υποχρεώνει να δεχθούμε παραπάνω εξουσίες. Το Ρήμι το δημιούργησαν πριν δημιουργηθεί, ε, κατά την, διαδικα... κατά την περίοδο κοίησης του οργανισμού. Είναι μια δύναμη αυτή που θα νικήσει τον εθνικό προστατευτισμό. Όλη αυτή η όθηση που μας δίδεται. Αυτά, Πρόεδρε, ίσως πάρω το λόγο μετά, αλλά ήθελα να σε γενικά θέματα και θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον ε, κύριο Διευθυντή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και φυσικά με τη βοήθεια των συναδέλφων μου. Κύριε Γιώργ, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα REMIT καταρχήν και το πλέγμα των δραστηριοτήτων που συνάπτονται με το πρόγραμμα αυτό. Όπως σας είπα, εμείς προετοιμάσουμε μια πιλωτική μελέτη με συμμετοχή διαφόρων ρυθμιστών για το πώς η εποπτεία της αγοράς βάσει του ρήμιτ θα μπορούσε να αναπτυχθεί και εξετάζουμε τι προκύπτει λοιπόν και τα διδάγματα τα οποία μπορούν να αντιληθούν για να επηρεάσουν και τις διαδικασίες μας. Εγώ βλέπω δύο τουλάχιστον διαστάσεις στο σημείο αυτό. Πρώτα απ' όλα να μπορούμε να έχουμε συνεργασία με την NRA, η οποία θα έχει εκτελεστικές και εφαρμοστικές εξουσίες, ενώ εμείς θα έχουμε αναλυτικές μονάχα. Ο στόχος μου λοιπόν είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τις εθνικές ρυθμιστικές ε, αρχές, NRAs, όταν υπάρχει πρόβλημα χειραγώγησης της αγοράς, υπό τη καταγγελόμενη χειραγώγησης, να παρεμβαίνουν και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην πυθό και όχι στην ε, εφαρμογή κυρώσεων. Να μπορούν λοιπόν οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν μια μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τη δράση τους. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε με μεγάλη, ε, με μεγάλη ταχύτητα τις εξελίξεις στην αγορά. Η πρόταση της Κομισιόν, και αυτό ήταν ένα στοιχείο που μας οδήγησε σε κάποιες ε, περαιτέρω ανησυχίες, ζητήθηκε να έχουμε 50 παραπάνω μέλη του προσωπικού, αλλά εγώ ε, μονάχα μπόρεσα να εμπλακώ σε ένα, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. 15 συγγνώμη και όχι 50 μέλη του προσωπικού είναι πολύ μικρός αριθμός και δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα, είχαν, θα είχαμε ανάγκη. Αν δούμε το αμερικανικό μοντέλο, Ξέρουμε ότι οι ρυθμιστές στις ΗΠΑ έχουν να αντιμετωπίσουν μια αγορά αντίστοιχη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητούμε μαζί τους για να δούμε τι ακριβώς είναι το επίπεδο, το σωστό επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Αλλά εγώ σκέφτομαι περισσότερο για 40 με 60 άτομα και όχι τα 15 που η Κομισιόν είχε διατυπώσει τότε στην πρότασή της είναι φανερό ότι εμείς θα χαιρετήσουμε οποιαδήποτε κίνηση προς ένα πιο συνεκτικό σύστημα καταγραφής για τους συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας σε όλη την ε, Ευρώπη, είτε παρέχουν ενέργεια είτε εμπορεύονται ενέργεια. Οποιαδήποτε κίνηση λοιπόν είναι θετική. Θα θέλαμε να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα σύστημα ενιαίου διαβατηρίου για τους φορείς στον τομέα της ενέργειας. Και τώρα σε ό,τι αφορά την εμπορία και τις συνδέσεις με τρίτες χώρες. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά για να μην δημιουργήσουμε παραθυράκια με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις ε, <clears throat> ρυθμίσεις μας ότι η εμπορία ενέργειας η οποία επηρεάζει την Ευρώπη άμεσα ή έμεσα να καλύπτεται από την εποπτεία που πρέπει εμείς να ασκούμε στον χώρο της αγοράς. Και αν τώρα μπορώ να περάσω στο θέμα της φιλελευθερωποίησης και τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με, την, ε, με τον ανταγωνισμό στον λιανικό τομέα ενέργειας. Αυτά τα θέματα είναι η αρμοδιότητα, η κοινή των εθνικών ρυθμιστών του δικού μας φορέα και της Κομισιόν. Η σωστή εφαρμογή του τρίτου πακέτου και η σωστή υλοποίηση αυτού του τρίτου πακέτου στην εθνική νομοθεσία είναι προφανώς κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσει προσεκτικά η Κομισιόν. Εμείς ως αποκεντρωμένος φορέας ασχολούμεθα περισσότερο με διαμεθοριακά θέματα, κυρίως στο επίπεδο χονδρικής, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο στο επίπεδο χονδρικής. Και φυσικά οι εθνικοί ρυθμιστές εξακολουθούν να διατηρούν ένα ρόλο και μία ε, ευθύνη σε ανεξάρτητο επίπεδο στις χώρες τους. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους εθνικούς εθνιστέ σε ορισμένε χώρες για να λάβουν υπόψη τους και να υποφελθούν από τις βέλτιστες πρακτικές. Μπορεί αυτό να μην σας φαίνεται πολύ συγκεκριμένο, αλλά ο φορέας μας είναι αυτός ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι θα λειτουργήσει καλά η εσωτερική αγορά και αυτή είναι μια κοινή αρμοδιότητα και κοινή μέρημνα όλων των θεσμικών οργάνων. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους εθνικούς ρυθμιστές και φυσικά έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κομισιόν για θέματα που είναι διαμοιραζόμενες αρμοδιότητες και θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και τώρα θα ήθελα... Θέλω να απαντήσω τώρα σε δύο παρατηρήσεις. Αναφέρθηκε το Ρήμιτ και πάλι. Φυσικά είναι μια μεγάλη πρόκληση για το φορέα μα γιατί αναλαμβάνει πραγματικά πολύπλοκες αρμοδιότητες ο φορέας μας, ο Acer. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι και μια πρόκληση για τους εθνικούς ρυθμιστές, γιατί μόνο πολύ λίγοι από αυτούς είχαν πραγματικά την ευθύνη της εποπτείας της εμπορίας ενέργειας. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν ικανότητες και τεχνογνωσία στο προσωπικό μας το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει μια σωστή συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν και της υπηρεσίας μας, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανές περιπτώσεις ε, χειραγώγησης ή κατάχρησης της αγοράς. Σίγουρα όμως το ρήμετ από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί θα ξεκινήσουμε εμείς την οργάνωσή μας και στον φορέα μας και να γίνει και η απαραίτητη συνεργασία των συντονιστών των ε, ρυθμιστών σε, συγγνώμη, σε εθνικό επίπεδο, γιατί πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις που εμπλέκουν δύο ή τρεις χώρες και πρέπει να υπάρξουν ομάδες ρυθμιστών που θα εξετάσουν κατά πόσο υπήρξε κάποιο πρόβλημα ή όχι. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και πιστεύω ότι το εκτενές πιλωτικό πρόγραμμα που κάναμε τους τελευταίους έξι περίπου μήνες μας έδωσε πολύ καλές ιδέες για το πώς πρέπει να οργανώσουμε τα θέματα αυτά, για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις από τη στιγμή που υπάρχει η πλήρης εφαρμογή αυτών των νομοθεσιών. Για το εμπόριο με τρίτες χώρες, το REMIT θα αντιμετωπίζει κάθε συναλλαγή που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει σημασία λοιπόν ποιο είναι ο ιδιοκτήτη ενέργεια ή ο εμπορευόμενος στην ενέργεια. Το REMIT όμως δεν μπορεί να αποφύγει προαιρέσει για την ε, γερμανική αγορά ενέργεια να την χάνουν εμπορία στη Σιγκαπούρη ή κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε όμως γίνεται στην αγορά τη στιγμία, την αγορά spot, θα καλύπτεται από το ρήμετ ανεξάρτητα από την ιδιότητα και την εθνικότητα των ιδιοκτητών και των εμπόρων. Υποδομές τώρα τι να πούμε για αυτό το θέμα. Όσον αφορά την υποδομή στον χώρο του φυσικού αερίου, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει το δίκτυο και βλέπουμε από τις ε, προσωμιώσεις που έχουν γίνει ότι εάν έχουμε... αν μπορέσουμε να οργανώσουμε σωστά την προσέγγιση θα μπορέσει το δίκτυο αυτό να μεταφέρει τους όγκους που απαιτούνται. Γι' αυτό δεν ε, χρειάζεται να δημιουργήσουμε επιπλέον ε, χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγών αερίου. Υπάρχει τέτοια ανάγκη για τον ηλεκτρισμό, όχι όμως για τους αγωγούς αερίου. Νομίζω ότι έτσι κάλυψα όλα τα θέματα. Επιτρέψτε μου να κλείσω ε, απαντώντας σε κάποια από τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Τούρμες. Τα χρήματα που έχουν διατεθεί για τις ε, υποδομές, όσον αφορά τα χρήματα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει επικάλυψη όσον αφορά τις πληρωμές. Αλλά θα πρέπει να θεσπίσουμε κριτήρια ώστε να κατανεμηθούν τα χρήματα αυτά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όσον αφορά ε, τις ε, ε δεν θέλω να δώσω την λάθος εντύπωση με τον νέο κανονισμό του από το 2010 έχει πιο ολοκληρωμένο ρόλο η Acer όσον αφορά την εποπτεία του μηχανισμού ε, και αυτός ο μηχανισμός μάλλον είναι ένα από τα βασικά συστατικά ώστε ε, να γίνει η σωστή αξιολόγηση των διασυνοριακών ε, εξελίξεων και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του πακέτου για τις υποδομές. Και τέλος, όσον αφορά την ανταπόκριση στη ζήτηση και, την, ε, και το σύστημα ε, διανομής. Ε, αυτά βρίσκονται στα άκρα των της αρμοδιότητάς μας, διότι εμείς ασχολούμαστε κυρίως με την χοντρική αγορά ενέργειας. Και αυτά τα θέματα δεν βρίσκονται ακριβώς στην καρδιά των αρμοδιοτήτων μας αλλά φυσικά συνομιλούμε με τους παραγόντες αυτούς, ε, γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό κομμάτι και όσον αφορά την ε, ανταπόκριση στη ζήτηση, στο βαθμό που αυτό έχει να κάνει με την ε, λειτουργία των συστημάτων, αυτά θα μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Όσον αφορά το 14 πρόγραμμα ανάπτυξης, δεν ξέρω αν πιο κατάλληλο χρονικό διάστημα είναι τα 10 ή τα 15 χρόνια. Νομίζω ότι τα 10 χρόνια είναι πολύ καλός τρόπος να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, και ε, πρέπει να δώσουμε τις ε, συστάσεις μας για τα θέματα αυτά και περιμένουμε αυτό το μήνα να έχουμε για την ένσοκτα τις μελέτες και την άλλη μελέτη τον άλλο μήνα. Πάντως πρόκειται για μία διαδικασία. Τα πηγαίνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και στο μέλλον θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Και όσον αφορά ε, τα διάφορα γεγονότα, νομίζω ότι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε να υπάρχει το σύστημα που θα για να αντιμετωπιστούν τα γεγονότα αυτά. Ε, όταν... Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει το σύστημα θα πρέπει η TSO να να φροντίσουν να μην υπάρχουν προβλήματα στην παροχή. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ευκαιρία αυτή να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σας. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας είναι ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποτότσνικ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπόλς και τον κύριο Μόγκ για το γεγονός ότι ήσασταν εδώ και ή μάλλον ξανά ήσασταν εδώ. Και φυσικά τα θέματα που συζητήσαμε εξακολουθούν ότι είναι στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Ακολουθεί το θέμα της ε, σύντομης έκθεσης του κυρίου Χάτζη Μαρκάκη για τις ε, συζητήσεις με το Συμβούλιο και τα θέματα κυριότητας και διαφάνειας της αγοράς εργασίας. Ήταν μια εργόδηση υπόθεση, αλλά έχετε το λόγο. Ναι, πράγματι το REMIT είναι το ακρονιμό για αυτό το σχέδιο. Μπορώ να σας πω ότι μαζί με πολλούς συναδέλφους έχουμε καταφέρει σε πρώτη ανάγνωση να εγκριθεί η οδηγία για το REMIT. Να σταθώ μονάχα σε μερικά σημεία τα οποία είναι σημαντικά για μας. Το πρώτο σημείο το έθεσε ήδη ο κύριος Ποτόσνικ και είναι το θέμα της καταγραφής όλων των εμπλεκομένων στον χώρο της ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο ελαφρό από ένα σύστημα αδειοδότησης. Επομένως, μπορούμε να έχουμε και μια λύση η οποία είναι και εθνική και ευρωπαϊκή για αυτούς οι οποίοι έχουν ευθύνη στον τομέα αυτό σε επίση στον τομέα της ε, εμπορίας αδειών εκπομπών και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα REMIT και αυτό είναι πολύ θετικό για την επιβολή κυρώσεων τώρα. Έχουμε συζητήσει για θέματα ενοποίησης, έχουμε συζητήσει απλώς τουλάχιστον να έχουμε κάποιους ελάχιστους κανόνες ώστε οι, τα πρόστιμα που επιβάλλονται να μπορούν να είναι ανάλογα με τη ζημία που υφίσταται ο καταναλωτής. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το έθεσε ο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κλώστ Τέρμις για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το, τη σχέση μεταξύ της Acer και των εθνικών ρυθμιστών, πρέπει να κάνω σαφές ότι ο διευθυντής που μόλις ε, γνωρίσαμε, τον κύριο Ποτόσνικ, θα έχει μια ενισχυμένη ανεξαρτησία ο διευθυντής της Acer. Αυτό θα κάνει κατά την άποψή μας και την ε, υπηρεσία Acer αλλά και το συνολικό σχέδιο Remit. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν ευρείες εξουσίες για την εφαρμογή του συστήματος Remit και επομένως υπάρχει μια ρήτρα μεταρρύθμισης ώστε στο μέλλον να μπορέσουν να διευρυνθούν αν χρειάζονται αυτές οι αρμοδιότητες. Για το θέμα της μορφής των εκτελεστικών μέτρων, εμείς θελήσαμε να ενισχύσουμε την εκτελεστική ικανότητα της ΕΣΕΣ στα θέματα αυτά. Επίσης, σε ό,τι αφορά το κείμενο, εμείς καταφέραμε να υπάρχουν πραγματικά οι ρυθμίσεις για κυρώσεις να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε σαφείς και απτές απώλειες οι οποίες πρέπει να τύχουν αποζημίωση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την ε, Ουγγρική Προεδρία με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί για τα θέματα αυτά. Μας έχει υποστηρίξει και η Κομισιόν φυσικά, αλλά η Ουγγρική Προεδρία έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργοκ ο οποίος και ο ίδιος έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ως Ούγγρος και βοήθησε να υπάρξει μια ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων και σε ψυχολογικό επίπεδο τα σημαντική παρουσία του και επίσης ο κύριος Τούρμες έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και μπόρεσε με ένα λυσιτελή τρόπο να προωθήσει τις ε, διαπραγματεύσεις οι οποίες χωρίς αυτό δεν θα είχαν καρποφορήσει τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι θα αποχωρήσω από την Επιτροπή Ενέργειας. Είναι η τελευταία μου εμφάνιση και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία του. τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά στο διάστημα αυτό και σας ευχαριστώ πολύ και για την ε, καλή και αξιόπιστη δουλειά που έχετε κάνει εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, συχνά είναι πολύπλοκη η δουλειά μας, θα σας δούμε όμως ε, κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα εκπροσωπείτε η πολιτική σας ομάδα από κάποιον άλλον στο μέλλον. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, ο Κλωτ Τούρμες έχει το λόγο. Πάντα μου φαίνεται ύποπτο όταν ακούω επένους για μένα. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα. και μου φαίνεται και ύποπτο ότι η Προεδρία λέει ότι έχει πετύχει πάρα πολλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εγώ είχα κάπως την εντύπωση ότι ήταν πολύ ήπιες οι διαπραγματεύσεις και ότι έχουμε εκχωρήσει πολλά στο Συμβούλιο. Ε, τώρα αυτό είναι μια πικρή σταγόνα στις, όλες τις ε, διαπραγματεύσεις. Παρουσιάσαμε μια σειρά ιδεών το θέμα της ε, καταχώρησης, αλλά τελικά την ε, ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το REMIT για να αναδιαρθρώσουμε ε, διαφορετικά την αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Νομίζω ότι Αυτήν δεν την εκμεταλλευτήκαμε επαρκώ. θα ήθελα περισσότερα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε μπροστά μα αυτό που έχουμε. ελπίζουμε η Acer να ε, αποκτήσει επαρκές προσωπικό και θα πρέπει να είναι ένα από τα καθήκοντά μας και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του χρόνου να φροντίσουμε Ε, να μπορέσει η Acer να εκτελέσει την αποστολή της και αυτό θα μπορέσει να το κάνει μόνο αν έχει επαρκές προσωπικό. Με αυτά τα, λίγα, τα λίγο πικρά λόγια... Ε, ελπίζω τελικά ε, η πρόταση αυτή να έχει ε, θετικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον πρόεδρο και όλους όσους συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Ο συνάδελφος Γκιούρκ. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μόνο για την ε, καλή δουλειά σας. Ο κύριος Τούρμες ήδη πήρε το λόγο και θα ήθελα και εγώ να γράψω την ευκαιρία να πω λίγα λόγια. Θέλω να σας καθησυχάσω, να σας ε, πω ότι είμαι πεπισμένος ότι μπορέσαμε να πετύχουμε το μέγιστο όσων μπορούσαμε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αναφέρατε μια σειρά θεμάτων ε, που θεωρείται σημαντικά. Δεν είναι όμως απαραίτητα εντός του πεδίου εφαρμογή ε, της αρχικής πρότασης. Μιλήσατε για την εισαγωγή νέων στοιχείων. Νομίζω ότι έχουμε ακολουθήσει τη σωστή προσέγγιση έχουμε ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση και έχουμε πετύχει ε, έναν συμβιβασμό και νομίζω ότι υπό τις συγκεκριμένε προϋποθέσεις αυτό ήταν το ε, βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Όλα έγιναν αρκετά γρήγορα, έχουμε όμως πολύ καλή ποιότητα νομοθετικέ διατάξει και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω γι' αυτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ήσασταν ε, πολύ αφοσιωμένο στο θέμα αυτό. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να το πετύχετε αυτό σε συνεργασία με την ε, Ουγγρική Προεδρία. Σα ευχαριστώ λοιπόν και είναι πραγματικά σπάνιο όλες οι ομάδες να είναι συγχρόνως ικανοποιημένες και το γεγονός ότι καταφέραμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα οποία διεκδικήσαμε, να τα προωθήσουμε και παρόλα αυτά η Προεδρία να είναι και αυτή ικανοποιημένη. Το βασικό είναι λοιπόν ότι περάσαμε όλα αυτά τα θέματα και το θέμα είναι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ και για αυτό το σημείο. Μπορώ να περάσω λοιπόν τώρα στο σημείο 7. Μάλλον τελείωσε το σημείο 7 και περνάμε στο σημείο 8 που είναι η έκθεση της κυρίας Κολάσκα Μπομπίνσκα και θα της δώσω ασμένος το λόγο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο ε, γνωμοδότησης για τις συλλογικές αγωγές έχει ένα χαρακτήρα συμβιβαστικό και νομίζω ότι πρέπει ως τιούτο να υποστηριχθεί από την Επιτροπή μας. Κάποιοι από εμά δεν θέλαμε να υπάρχουν συλλογικέ πρόσφυγες με τη λογική ότι αυτό θα άνοιγε το δρόμο για καταχρηστικού ε, χαρακτήρα δικαστικές διαδικασίες. Εγώ αντίθετα θεωρώ ότι η συλλογή προσφυγή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Η... Τα θετικά στοιχεία λοιπόν αυτού του συστήματος για τους πολίτες υπερκεράζουν τα αρνητικά στοιχεία πιθανών καταχρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα ευρωπαϊκού χαρακτήρα σύστημα για τα θέματα συλλογικής προσφύγης. Συγχρόνως χρειαζόμαστε ε, κάποιες διασφαλίσεις για να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις εναντί τέτοιων προσφύγων. Θέλουμε να έχουμε σαφείς κανόνες για την αστική ευθύνη, τη δοσηδικία και το, ε, το παραδεκτό τέτοιων δράσεων. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σαφείς κανόνες για το τι είδους προσφυγές μπορούν να είναι αποδεκτές. Παραδείγματος χάρη όρια για το ποιοι μη κυβερνητικοί φορείς και εθνικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες προσφυγές. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση από την πλευρά αυτών οι οποίοι αναλαμβάνουν μια προσφυγή ότι αν υπάρξει αρνητική απόφαση θα μπορούν να επομιστούν το κόστος το δικαστικό. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες δοσηδικίας. Δεν πρέπει να υπάρχει επιλογή δικαστικών ε, ε, δικαστικών χώρων προσφυγής που να επιλέγουν αυτοί οι οποίοι καταθέτουν μια προσφυγή το καλύτερο κράτος μέλος για να ευδοκιμήσει η προσφυγή τους. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Δεν μπορούμε φυσικά ποτέ να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν υπόκειται σε καταχρήσεις, αλλά οι διαφυλάξει που θα πρέπει να θεσπίσουμε θα πρέπει να αποτρέψουν τις ακρότητες του Αμερικανικού Συστήματος Συλλογικών Προσφυγών που πάντα παρουσιάζεται σε ένα σύστημα το οποίο οδηγεί σε καταχρήσει. Και οι εταιρείε αλλά και οι καταναλωτέ θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται και στα δικαιώματα αλλά και στι ευθύνε. Κάποιοι από του συναδέλφους μα θέλαν να προωθήσουν ακόμα περισσότερο το σύστημα αυτό με την πλήρη εναρμόνιση των συστημάτων συλλογική προσφυγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμφωνώ με μια τέτοια οδηγογραμμή αλλά δεν νομίζω ότι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι τα νομικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρουν παρασάγκας το ένα από τα άλλα. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα το οποίο θα είναι κοινό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα βασίζεται σε ελάχιστες προδιαγραφές και η Κομισιόν θα πρέπει να μας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα διέπουν τα περαιτέρω μέτρα τα οποία μπορούν να θεσπίσουν τα κράτη-μέλη προαιρετικά, εάν το επιθυμούν. Έτσι σεβόμεθα για την αρχή της επικουρικότητας και δίνουμε και μια βασική προστασία σε όλους τους καταναλωτές όπου και να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, το σύστημα συλλογικής προσφύγης θα πρέπει να βελτιώσει και να διευκολύνει την πρόσβαση στα δικαστήρια, αλλά και οι, εναλλακτικοί, οι μηχανισμοί εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί να είναι πολύ πιο ταχύς και λιγότερο δαπανήρη. Επομένως, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του μηχανισμού αντιμετώπισης και επίλυσης διαφορών που θέλουν να ακολουθήσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν και προσβλέπω στις τροπολογίες που θα πρέπει να καταθέσουν οι συνάδελφοι μέχρι την, μέχρι την Πέμπτη. Ευχαριστώ κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ε, Πικροτώ την έκθεση της κυρίας Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Νομίζω ότι είναι ε, πολύ σαφής, ε, πολύ πλήρης και πολύ αναλυτική. Έχει ε, ιδιαίτερα καλή διατύπωση όσον αφορά τα διάφορα εχέγγυα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα πράγμα που μου αρέσει ιδιαίτερα. Το θέμα του περιορισμού των κριτηρίων των φορέων που μπορούν να συμμετέχουν. Διότι δεν νομίζω ότι θέλουμε να βρεθούμε ε, στην κατάσταση να δημιουργηθεί ολόκληρη βιομηχανία ε, όπως, ε, αντιδικιών όπως ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενδεχομένως θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τρόπος να το κάνουμε αυτό θα ήταν να περιοριστούμε σε αυτούς ε, που έχουν θυγεί από την δράση ή αυτούς ε, που έχουν ε, ένομο συμφέρον, ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία σχετικής βιομηχανίας. Για τρία σημεία θα μπορούσα να υποβάλω τροπολογίες για να αναπτύξω λίγο τα θέματα αυτά. Μία ομάδα ανθρώπων που θα μπορέσουν να ωφεληθούν ιδιαίτερα από ε, τις ε, συλλογικές προσφυγές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι δεν έχουν τους πόρους ε, να αναλάβουν δράση απέναντι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη ε, της μείωσης ε, του κόστους ε, και να είναι όσο γίνεται πιο απλές τις σχετικές διαδικασίες. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Κομισιόν να υποβάλει κάποιες καινοτόμες λύσεις για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν θέλουν να προσφύγουν ώστε να η ε, δυνατότητα που δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να ε, προσφύγουν να μην είναι απλά θεωρητικές. Δεύτερον, θα ήθελα οι συλλογικές προσφυγές να περιλαμβάνουν και το περιβαλλοντικό δίκαιο, διότι συχνά έχουμε την περίπτωση όπου άτομα και επιχειρήσεις επηρεάζονται από κάποια περίπτωση ρήπανσης που ξεπερνάει ε, τα σύνορα μιας χώρας. Ε, είχαμε πέρσι το φθινόπωρο ε, μια περίπτωση με την Ουγγαρία και την ρήπανση του Δούναβη. Θα ήθελα εδώ να σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι δυνατή η συλλογική προσφύγη, διότι εδώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί πολύ καλά η αρχή ο, ιτόμενος, ο, πληρώνει. Και ε, τίθεται το θέμα του αν ε, στις συλλογικέ ε, προσφυγέ θα πρέπει να ισχύει το opt-in ή το opt-out. Η ρήτρα προαιρετικής ρητρα προαιρετικη συμμετοχη η ρήτρα μη συμμετοχή. Και δεν ξέρω ποια θα ήταν η καλύτερη λύση, διότι ενώ σε πολλέ περιπτώσει η ρήτρα προαιρετική συμμετοχή να είναι καλύτερη, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει όπου η ρήτρα προαιρετική μη συμμετοχή είναι ο μόνο τρόπο να ε, διασφαλιστεί η δυνατότητα σε όλους ε, να προσφύγουν. Διότι κάθε μεμονωμένη προσφυγή θα ε, είναι μικρής αξίας, αλλά θα έχουμε μεγάλη ομάδα ανθρώπων που έχουν φυγεί. Για παράδειγμα, ένα ελαττωματικό προϊόν και μπορεί πολλοί καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη να έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Θα είναι όμως ε, δύσκολο να οργανώσει κανείς ε, τη συλλογική προσφυγή και συμφωνώ ότι η πληροφόρηση σε τέτοιες περιπτώσεις ε, θα είναι πολύ σημαντική. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Πάντως θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της αυτή. Ευχαριστώ. Τη γνωμοδότηση, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Όπως είπε και η κυρία Κολάσκα Μπομπίσκα, την Πέμπτη είναι κατα... Ε, καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες, ο κύριος Τούρμες και η Κομισιόν. Ο Κλοντ πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Λένα για την τόσο ισορροπημένη αυτή έκθεση. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη υποστήριξη στην πολιτική σου ομάδα για τις συλλογικές προσφυγές και ως εκ τούτου έχει επιτύχει μια ισορροπία η οποία δεν ήταν και τόσο εύκολη. Ένα θέμα για το οποίο εμείς θα πρέπει να έχουμε σαφήνεια είναι το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τα οποία αναμένουμε από την Κομισιόν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν νομοθεσία πλαίσιο, ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι προτιμούν μια τομεακή, μια κατατομής προσέγγιση. Το πρόβλημα με μια νομοθεσίας πλαίσιο είναι ότι θα είναι τόσο αχανής ώστε να μην αντιμετωπίζει αρκετά λεπτομεριακά τις ανάγκες των διαφόρων τομέων. Και μετά από τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε ως σκιώδες εισηγητές, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί σου και να συζητήσουμε ποια είναι η άποψή μας για αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, ότι χρειάζεται ορισμένες φορές να υπάρχει για τους καταναλωτές, για τον ανταγωνισμό, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μία κατά του περιβάλλοντος, συγγνώμη, μία κατατομής προσέγγιση και ειδική λεπτομεριακή νομοθεσία για να έχουμε καλύτερα στοχευμένα εργαλεία. <clears throat> Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες σε σχέση με τη διαδικασία δύο σταδίων για τις δοκιμαστικές περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ορισμένε από τι επικρίσει που έχουν διατυπωθεί. Τι είναι αυτή η διαδικασία στη χώρα η οποία επηρεάζεται περισσότερο θα πήγαινε κανείς στο δικαστήριο και θα καθόριζε θα, την κατανομή των ευθυνών. Αυτό θα είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη φάση θα ήταν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, οι φορείς από άλλες χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πρώτη απόφαση <clears throat> και να την επικαλεστούν για να ζητήσουν αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει υποστηριχθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο του Παρισιού και από, τον, ε, από την Ένωση των Δικηγόρων στο Βερολίνο και έχει την υποστήριξη λοιπόν της γαλλικής ε, ε, Γερουσίας και του γερμανικού Bundesrat που είναι το αντίστοιχό της. Έχουμε λοιπόν μια ευρύτατη υποστήριξη για μια τέτοια διαδικασία στις μεγάλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σωστό βέβαια το ότι τονίστε το κίνδυνο να υπάρξει κάποια να υπάρχει διαδικασία επιλογής των δικαστικών ε, χώρων να διαλέγει κανείς το πιο πρόσφορο χώρο. Και αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν τώρα άλλοι τομείς όπου εμείς έχουμε ισχυρές αντιρρήσεις με την ε, έκθεσή σας γιατί περιέχει, τη γνωμοδότηση, περιέχει και την αρχή ο ιτόμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα. Το θέμα είναι ότι όπως είπε και η Φιώνα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη έχουν πρόβλημα για να πληρώσουν τους δικηγόρους τους. Από την άλλη μεριά έχετε μια μεγάλη επιχείρηση η οποία μπορεί να αγοράσει, μάλλον μπορεί να προσλάβει 5, 8, 10, 50 δικηγόρους. Εάν τώρα η αρχή είναι ότι ο ιτόμενος στη δίκη πληρώνει το νομικό κόστος, το δικαστικό κόστος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις <clears throat> μόνο ακούγοντας ότι πηγαίνει στο δικαστήριο ο αντίπαλός τους με 15 δικηγόρους και φαίνει και μερικούς τεξανούς δικηγόρους που είναι ακόμα πιο ακριβοί, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ υψηλό το τίμημα μιας ήτας στο δικαστήριο βάσει της αρχής του ότι ο ιτόμενος πληρώνει τα δικαστικά έξοδα. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα τεράστιο φράγμα, ένα τεράστιο εμπόδιο για τις οργανώσεις πολιτών και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να φέρουν τα πράγματα αυτά στο δικαστήριο. Χρειάζεται λοιπόν εδώ μια λύση ή δεν θα πρέπει να αναφέρουμε καθόλου το θέμα αυτό και από ό,τι μου είπανε Υπάρχει ένας κανονισμός για τις ε, δίκες για μικροποσά, για μικροϋποθέσεις που καλύπτονται από ένα κανονισμό και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε αν αυτός ο κανονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα ώστε να μην είναι αποτρεπτικό το πρόβλημα του δικαστικών, δικαστικών εξόδων για τους διαδίκους. Έχουμε καταθέσει λοιπόν μια, ένα μικρό αριθμό από τροπολογίες και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σου και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή λύση για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια ήδη είχε έρθει ενώπιον μας το θέμα των συλλογικών προσφυγών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει την ιδέα αυτή. Και πρέπει και πάλι να αναφέρω τις ανησυχίες που τρέφω για το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι θα μπλέξουμε <clears throat> και δεν ξέρω ότι αν, μπλέξουμε σε ένα τέτοιο σύστημα μέχρι που θα φτάσουμε. Δεν ξέρω. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει μια εισβολή του αγγλοσαξονικού δικαίου στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Κατανοώ ότι η συγγήτρια θέλει να συμπεριλάβει στη γνωμοδότησή της και κάποιες διαφυλάξεις. Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο γιατί εάν δεχτούμε <clears throat> αυτές τις συλλογικές προσφυγές θα πρέπει να έχουμε διαφυλάξει. Αλλά πρέπει να έχουμε συλλογικές ε, προσφυγές. Έχω την εντύπωση ότι ανοίγει το κουτί της πανδώρας η Κομισιόν. Με αυτό το μέτρο. Και δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο θετικές οι συνέπειες όπως αυτές που περιέγραψε η συγγήτρια, οι συνέπειες για τον καταναλωτή, οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Ο φόβος μου είναι ότι ανοίγοντας τους ασκούς του αιώλου θα έχουμε σοβαρές συνέπειες οι οποίες θα εμφανιστούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μου λέτε ότι είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξη για το θέμα αυτό. Μπορεί. Αλλά δεν μπορώ παρά μόνο να σας αναφέρω τις βαθιές ανησυχίες που έχω. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κάπως πρόωρα το να θεσπίσουμε τέτοιους μηχανισμούς μέσα στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο τη στιγμή που έχουμε τους εθνικούς δικαιακούς χώρους δεν νομίζω ότι έχουμε πράγματι συνυπολογίσει τις συνέπειες και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτό το μέτρο. Έχουν αναφερθεί βέβαια οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Εγώ παρακολούθησα όλο αυτό το θέμα πολύ προσεκτικά και πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ τα μάλα και δεν θα ήθελα να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό του, των συλλογικών προσφυγών. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε, ναι, αλλά θα πρέπει να το θέσουμε στο σωστό πλαίσιο και με τέτοιες διαφυλάξεις, ώστε μετά από μερικά χρόνια να μην κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας ότι έχουμε πράγματι δημιουργήσει μια ορολογιακή βόμβα. Σας ευχαριστώ και ρωτώ αν η Κομισιόν θέλει να παρέμβει. Αν όχι, να δώσω το λόγο στην κυρία Κολοσκοποπίνσκα σύντομα. Α, η Κομισιόν, παρακαλώ. Μόνο θα πρέπει να βιαστούμε λίγο. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την ε, τελευταία φορά που βρέθηκα στην Επιτροπή σας υποσχέθηκα ότι θα επανέλθω με τα αποτελέσματα της ε, δημόσιας διαβούλευσης που δεν μπορούσα να σας δώσω κατά την προηγούμενη συνεδρίαση λόγω του τεράστιου όγκου απαντήσεων και πράγματι έχουμε λάβει πάνω από 300 απαντήσεις από διάφορους ενδιαφερομένους, ε, από ενώσεις επιχειρήσεων, ε, εκπροσώπους των καταναλωτών και άλλων. 14 ε, από τα 27 κράτη-μέλη επίσης απάντησαν, το οποίο δεν σημαίνει συχνά, και έχουμε λάβει επίσης περίπου 20.000 επιστολές από πολίτες. Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι επικροτούν την προσπάθεια να βρεθούν κοινέ αρχές για τις συλλογικές προσφυγές ακολουθώντας την προσπάθεια να βρεθούν αρχές ε, για τον κάθε τομέα δικαίου που θα εφαρμόσετε στην κάθε περίπτωση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ε, τώρα, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Ο κόσμος ε, τονίζει την ανάγκη εξέβρεση επαρκών εχέγγυων κατά των καταχρηστικών προσφυγών. Στο πλαίσιο αυτό, αυτό που ακούμε πιο συχνά είναι αφενός αναφορά στις ε, αμερικανικού τύπου συλλογικές προσφυγές, πράγμα που θέλουμε να αποφύγουμε ε, με κάθε τίμημα. Και επίσης στο πλαίσιο αυτό, ε, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προτιμούν το opt-in παρά το opt-out, τη ρήτρα προαιρετική συμμετοχής και όχι μη συμμετοχή. Επίση, ω κοινή αρχή υπάρχει αίτημα από του ενδιαφερομένου να προωθηθεί η εναλλακτική επίλυση διαφορών, η οποία κατά προτίμηση δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Να υπάρχει δηλαδή ε, προαιρετικός μηχανισμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για να μπορεί να ξεφύγει κανείς από την ε, δυνατότητα ε, δικαστικής συλλογικής προσφυγής. Η εικόνα όσον αφορά την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ενεργήσει πέρα ε, από το θέμα των κοινών αρχών ε, δεν είναι πολύ σαφής. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ανάγκη, της Ευρωπαϊκής Ένωση, την, ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει δεσμευτικά μέτρα, βλέπουμε ότι είναι υπέρμενοι οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, είναι κατά όμως οι ενώσεις επιχειρήσεων, ενώ τα κράτη-μέλη... μερικά συμφωνούν και μερικά διαφωνούν. Επίσης, το αποτέλεσμα της ε, δημόσιας Διαβούλευση δείχνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θέλουν ε, ο μηχανισμό συλλογικών προσφυγών να ισχύει όχι μόνο για τους καταναλωτές ε, όταν είναι θύματα, αλλά και για τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ισχύει ο μηχανισμός αυτός. Και το τελευταίο πράγμα που μπορώ να αναφέρω είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι πιστεύουν ε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, οντότητες που να εκπροσωπούν είτε το γενικό συμφέρον είτε ε, τα άτομα που εκπροσωπούν. Υπάρχει όμως εδώ διαφωνία εάν αυτές οι οντότητες θα πρέπει να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Νομίζω ότι το βασικό μάθημα εδώ είναι ότι η προσπάθειά μας είναι σημαντική και ότι δεν έχουμε σαφή κατεύθυνση ε, από, με, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ε, ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τις βασικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κολάσκα από Πίνσκα. Όπως βλέπουμε υπάρχουν ε, διστάμενα συμφέροντα ε, διότι από τη μία μεριά έχουμε τους καταναλωτές, από την άλλη μεριά όμως έχουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες φοβούνται πολύ τις καταχρηστικές προσφυγές και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τις αποφάσεις που θα λάβουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εφιώνα, η οποία έφυγε μεν, ναι, ανέφερε όμως το ειδικό ταμείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει η Κομισιόν για να βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσφεύγουν κατά μεγάλων επιχειρήσεων. Εγώ θα ήμουν κατά μια τέτοια δυνατότητα, διότι ήδη έχουμε σημαντικά προβλήματα με τον προπολογισμό. Το να δημιουργήσουμε ειδικό ταμείο για να στηρίξουμε αυτού που θέλουν να ασκήσουν ε, ε, δίωξη, αυτό θα είναι δύσκολο. Διότι τότε μπορεί να υπάρξει κατάχρηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιε ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει που δεν έχουν επαρκή πόρου για κάτι τέτοιο και ότι θα είναι δύσκολο για αυτού, αλλά το να τους δώσουμε οικονομικά τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγέ, νομίζω ότι αυτό είναι τρόπο να του βοηθάμε να καταχραστούν το σύστημα. Ε, δεν είναι, πρόκειται πάντα για μικρές επιχειρήσεις κατά μεγάλων. Ε, ε, συχνά είναι μικρές επιχειρήσεις που προσφέρουν κατά μικρών επιχειρήσεων. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστή λύση αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και ίσως θα πρέπει να υποστηρίξουμε πιο ένθερμα την εναλλακτική διευθέτηση διαφορών. Είναι προτιμότερο πάντα παρά η νομική λύση. Ε, ίσως να μην τονίζεται αρκετά όσο πρέπει στην γνωμοδότησή μου. Αλλά είναι ο τρίτος δρόμος όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλη ε, όλες οι εναλλακτικές μέθοδοι επιλύσεως των διαφορών και μπορούμε να έχουμε αυτό το σύστημα με δύο φάσεις, Κλοντ. Αντί να έχουμε το σύστημα επίπεδο χώρας μετά επίπεδο που είναι πάνω από τη χώρα, να έχουμε την εναλλακτική ε, ρύθμιση των διαφορών, διαθέσει διαφορών σε μία φάση και μια άλλη λύση θα είναι η λύση δικαστική, νομική. δεύτερη προσοχή. Περιμένω τις τροπολογίες και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε ένα-δύο πράγματα και θα χαιρόμουν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας αποστείλει τα αποτελέσματα της συζητήσεως, τη σύνοψη των διαβουλέψεων που αναφέρατε. Θα μας βοηθούσε κάτι τέτοιο πριν λάβουμε τελική απόφαση. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κάτι τελικό όσον αφορά τις συζητήσεις και το τελικό αποτέλεσμα, ίσως όμως να είναι κάποιες ιδέες, κάποιες ερωτήσεις, κάποια πράγματα που αναφέρθηκαν που να μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ. Okay.